Καλησπέρα σας. Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε τις συνεδρίες της Επιτροπής μας. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Καλησπέρα σας. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίας επιτροπής μας που προβλέπεται από τις 3 μέχρι τις 6.30. Θα ήθελα πρώτα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξή μας. Αν δεν έχετε αντίρρηση, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 30ης και 31ης Μαρτίου 2015 και 6 και 7ης Μαΐου 2015. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις ε, μέχρι το τέλος συνεδρίασης, θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένα τα πρακτικά. Περάμε στο σημείο 3 τώρα. ανακοινώσει της Προέδρου. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι μετά από αίτημα της κυρίας Μορβάη να λάβει μέρος σε μια αποστολή της Επιτροπής ε, Γυναικών στην Ιρλανδία 24 και 25 Σεπτεμβρίου του 2015 η κυρία Μορβάη ζήτησε να μεταβεί εκτός ποσόστοσης με βάση το άρθρο 4.1β και ακολούθησε γραπτή διαδικασία μεταξύ των συντονιστών προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο θα δοθεί ε, η συμπερίληψη της κυρίας Μορβάη στην αντιπροσωπεία. Η πλειοψηφία των συντονιστών της Επιτροπής Γυναικών ήταν κατά της ε, έγκρισης αυτού του αιτήματος της κυρίας Μορβάη. Αυτή είναι η σύσταση των συντονιστών. Να μην γίνει δεκτό το αίτημα της κυρίας Μορβάη. Έχετε παρατηρήσει σχετικά. Δεύτερη ανακοίνωση. Στις 26 ε, Μαΐου είχαμε μια τριμελή αντιπροσωπεία της Επιτροπής Γυναικών που μετέβει στη Γενέβη. Η αντιπροσωπεία μας απαρτιζόταν από εισηγητές ε, της Επιτροπής ε, για την έκθεση ισότητας ε, των δύο φύλων και χειραφέτηση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή. Η συγγήτρια Τέρι Ρέντ ζήτησε να της δώσω το λόγο για να μας ενημερώσει για το τι συνέβη στην αντιπροσωπή αυτή, πώς εξελιχθεί η εργασία. Τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ήθελα μόνο εν συντομία να σας παρουσιάσω τα όσα εξετάσαμε κατά τη διάρκεια της αντιπροσωπείας αυτής. Ήμουν και εγώ και η Τζούλι Βόρτα από τους Σοσιαλιστές και η Καθρίν Βιέρα από την Άλντε. Forum, Visas Forum, το οποίο εξετάζει ευρύ φάσμα θεμάτων, ε, τεχνολογίες πληροφορικής, κοινωνίας πληροφορίας και το καθεξής, ITU, UNESCO, UNTA και ITI Women. Και ένα από τα ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί ήταν και το θέμα της ισότητας μεταξύ των φύλων. Ξέρετε ότι θα έχουμε μία έκθεση πρωτοβουλία για τις γυναίκες στην ψηφιακή εποχή και θέλαμε να διερευνήσουμε τι έχουν κάνει τα Ηνωμένα Έθνη σε αυτό το πεδίο. Γιατί έχει γίνει δουλειά και έχουν γίνει και διάφορε προτάσεις. Είχαμε πολύ ωφέλιμες ε, συναντήσεις με εκπροσώπους ε, του επιχειρηματικού κόσμου, ακτιβιστριών, επιμέρους ε, οργανώσεων του ΟΗΕ και συνοπτικά σε αυτό το ζήτημα υπήρξε μεγάλη έμφαση στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευση σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό αλφαβητισμό λοιπόν των γυναικών και την πρόσβασή τους στα ψηφιακά μέσα. Είναι ένα από τα θέματα που κατά τη γνώμη μου θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον να εξετάσουμε και στην έκθεσή μας. Όμως μαζί με αυτές τις προτεραιότητες Νομίζω ότι όλα τα μέλη της ε, αντιπροσωπείας θεώρησαν ότι πρέπει να διαβρύνουμε κάπως ε, το πεδίο αυτό. Τα ζητήματα λοιπόν τα οποία έχουμε εντοπίσει κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αφορούσαν και τη χρηματοδότηση, ποια προγράμματα και καθεστώτα προγραμμα... χρηματοδότηση μπορούν να αξιοποιήσουν οι γυναίκες εάν θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον τομέα, της ε, ίσης πληρωμής στον τομέα της πληροφορικής, γιατί υπάρχουν τεράστιες ανισορροπίες στις απολαβές ανδρών και γυναικών, μετά και πάλι το θέμα των ποσοστώσεων. Αν δείτε και τα στοιχεία, ιδίω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εκπροσώπηση ε, των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων πληροφορική είναι μεταξύ 4 και 7%. Θα πρέπει λοιπόν να το διαρευνήσουμε περαιτέρω. Και μετά και το ζήτημα τη βία κατά των γυναικών, παρενόχληση μέσω διαδικτύου, είναι σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε. Μετά συνάντηση που είχαμε με εκπρόσωπο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για την ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας και πώς ε, ε, αυτή επηρεάζει τις γυναίκες. Όλα αυτά τα θέματα μπορούμε να και πρέπει να τα εξετάσουμε στο πλαίσιο της ε, έκθεση ίδια πρωτοβουλία. Νομίζουμε ότι αυτή η αντιπροσωπή ήταν πολύ σημαντική και χρήσιμη για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Τώρα, στα πλήν στα αρνητικά αυτού του φόρουμ, παρότι συναντηθήκαμε με πολύ δραστήριες και δυναμικές γυναίκες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Όμως, ε, στις εναρκτήριες ομιλίες, νομίζω ήταν 12 μέλη ε, του πάνελ και όλοι ήταν άντρες. Και αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε περαιτέρω τις γυναίκες, ιδίω σε αυτό τον τομέα. Και εμείς ως Επιτροπή Γυναικών θα πρέπει ε, να ασκήσουμε πιέσεις, να προβάλλουμε περισσότερο αυτό το θέμα. Νομίζω ότι καμία από τις δύο συναδέλφους ε, δεν είναι εδώ για να πει κάτι παραπάνω, όμως αν έχετε ερωτήματα, αν κάτι άλλο συμβαίνει στις ομάδες σας, αν έχετε συζητήσεις, εκδηλώσεις για αυτά τα θέματα, μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μου γιατί με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ρέντ. Θέλει άλλος κανείς το λόγο, κυρίως ε, αν ε, είχαν, αν είχε λάβει μέλο στην αντιπροσωπεία. Αλλά απουσιάζουν οι άλλε ε, δύο συνάδελφοι που είχαν μεταβεί στη Γενέβη. Εν πάση περιπτώσει, για να ολοκληρώσω αυτό το σημείο με τι ανακοινώσει θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι σε ό,τι αφορά τη διαδικασία υποβολής των ε, για τον προϋπολογισμό του 2016, οι συντονιστές ε, στη συνεδρίαση της 16ης Μαΐου αποφάσισαν να ψηφίσουν τις τροπολογίες στον προϋπολογισμό στη συνεδρίαση της 13ης και 14ης Ιουλίου. Περνάμε τώρα στο σημείο 4 της ημέρης της διάταξης που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων για το θέμα των γυναικών που εργάζονται σε οικιακές εργασίες ε, ε, ή φροντίζουν ε, ε, άλλα μέλη της οικογένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγγήτριά μας είναι η κυρία Κωνσταντίνα Κούνεβα, στην ευρωπαικη ενωση η συγκεκρια μας ειναι η κυρια κωνσταντινα κουνεβα στην οποια θα δώσω και το λόγο για να μας παρουσιάσει το σχέδιο εκθεσής της. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες πρώτες σκέψεις και θα ήθελα να ακούσω τις αντιδράσεις σας και τις δικές σας ιδέες ώστε να καταλήξω σε ένα κείμενο το οποίο θα περιλαμβάνει όσες περισσότερες γίνεται από τις ιδέες όλων μας ώστε να καταλήξουμε στις διάφορες πλευρές του θέματος όσο πληρέστερα γίνεται. Να θυμίσω πως εμείς είμαστε συνεργαζόμενη επιτροπή στο θέμα των απασχολούμενων γυναικών ως οικιακών βοηθών με την Επιτροπή Απασχόλησης η Επιτροπή απασχόληση είναι αρμόδια για θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση της Διεθνού Οργανώση εργασία. Η Επιτροπή Απασχόληση θα ε, ασχοληθεί με τον αν η σύμβαση έχει κυρωθεί, πώς έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, αν εφαρμόζεται, αν υπάρχουν νόμιμα συμβόλαια κτλ. Εμείς θα επικεντρωθούμε περισσότερα σε άλλα θέματα όπως τα παρακάτω. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν τις γυναίκες στην οικιακή εργασία. Μήπως υποκατιστά φροντίδες που παλιά παρήχαν οι γυναίκες που έμεναν στο σπίτι. Μήπως σημαίνει πως η φροντίδα για άτομα μέσα στο σπίτι εξακολουθεί ακόμα να θεωρείται γυναικεία υπόθεση πρέπει να δούμε πώς παρέχονται οι υπηρεσίες π.χ. για παιδιά ή για ηλικιωμένους από κράτη που έχουν τις σχετικές υποδομές. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του βορρά και του νότου της Ευρώπης. Ποιες είναι οι καλές πρακτικές. Τι και να υπάρχουν σε, όλες, σε άλλες χώρες. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Τελείως ενδεικτικά να αναφέρω την πρακτική με τα κοπόνια μέσα νόμιμων εταιριών που σε χώρες όπως το Βέλγιο λειτουργούν με απόλυτη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Πρέπει να μας απασχοληθεί το ζήτημα του μεγάλου αριθμού των μεταναστριών που απασχολούνται στον τομέα της οικιακής εργασίας. Μπορούμε πλέον να μιλάμε για τελικοποίηση των μεταναστευτικών ρευμάτων διότι οι γυναίκες μετανάστρες είναι πιο εύκολο να βρουν τέτοιες δουλειές προκειμένου όμως να διασφαλίσουν την επιβίωση της οικογένειάς τους πέφτουν στην παγίδα πως θα δουλέψουν λίγα ακόμα και λίγα ακόμα και τελικά πακεντεύονται σε τέτοιες μορφές άτυπης απασχόλησης. Τα χρόνια περνούν χωρίς να είναι επαρκώς καλυμμένες ώστε να το, για το διάστημα που δουλεύουν αλλά και χωρίς να έχουν διασφαλίσει δικαιώματα συνταξιοδότησης. Μιλάμε περίπου για ζωές χαμένες. Βεβαίως όλα αυτά συμβαίνουν διότι υπάρχουν μεγάλα νομικά κενά ως προς την ρύθμιση αυτών των επαγγελμάτων Κάποιες χώρες έχουν προσπαθήσει να ρυθμίσουν τα ζητήματα με διαφορετικούς τρόπους, αλλά βρισκόμαστε ακόμα μακριά από ένα ενιαίο πλαίσιο που θέτει κοινέ αρχές. Αρχές που διασφαλίζουν το σεβασμό και τα δικαιώματα των εργαζομένων που τους επιτρέπουν να έχουν μια κοινωνική ζωή στο φως και μια αξιοπρεπή συνταξιοδότηση. Αυτό που θα πρέπει επίσης να ερευνήσουμε είναι κατά πόσο ακόμη και αν το επάγγελμα των οικιακών βοητών είναι ρυθμισμένο σε κάποιες χώρες μήπως αφήνει περιτόρια παραβιάσεων. Να αναφέρω ενδεικτικά το θέμα των μονοπροσώπων εταιριών αυτοαποσχολούμενων στη Γερμανία που δεν είναι σαφές με ποιο τρόπο υποχρεούνται στην παροχή κοινωνικής προστασίας. Η εκπαίδευση και αυτοπροστασία πρέπει επίσης να μας απασχολεί. Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν χωρίς να είναι πουθενά δηλωμένοι δεν έχουν και καμία πρόσβαση σε εκπαίδευση όσον αφορά την απασχόλησή τους. Η οικιακή εργασία όμως δουλεύουν συχνά σε συνθήκες αντιγυηνής και απαιτούν ειδικέ γνώσει και ειδικού κανόνες προστασίας. Πώ θα προστατεύσουμε αυτές τι γυναίκε, Χρειάζεται οργάνωση και συσπήρωση. συνήθω οι ομοσπονδίε εργαζομένων δεν απασχολούνται με αυτού του τομεί τη εργασία. Η κοινή οργάνωση όμω θα φέρει αυτέ τι γυναίκε στην επιφάνεια. Θα του δώσει φωνή και μεγάλη δύναμη θα τις απλάσει, από πολλούς φόβους. Πρέπει να βοηθήσουμε στην προσέγγιση τους από τα συνδικάτα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να επισημάνω στο τέλος είναι πως άσχεται από τα αίτια εργασία εντός σπιτιού ζητάτε από γυναίκες σε άλλες γυναίκες. Ζητάτε δηλαδή από γυναίκες που έχουν τα μέσα να πληρώσουν άλλες γυναίκες για να τους κάνουν τη δουλειά. Αυτό για μένα σημαίνει κάτι εξαιρετικά σημαντικό το οποίο ίσως δεν έχει γίνει επαρκώς κατανοητό ώστε από εμάς τις ίδιες. Όταν άλλες γυναίκες δουλεύουν για εμάς, μας επιτρέπουν να συνεχίζουμε αδιάσπαστα τη ζωή μας, την καριέρα μας, την κοινωνική μας ζωή. Έχουμε σκεφτεί πραγματικά πως όταν αυτές οι γυναίκες δουλεύουν χωρίς ασφάλιση και δικαιώματα θυσιάζουν τη δική τους ζωή και τη δική μας. Ένα σχόλιο που σοκάρει είναι η έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ γυναικών. Έχουμε λοιπόν και εμείς μεγάλο μερίδιο ευθύνης στο να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες οικιακά εργαζόμενες έχουν όλα τα δικαιώματα που τους εξασφαλίζουν μια αξιοπρεπή ζωή με την απαραίτητη ασφάλιση και προστασία και μια αξιοπρεπή συνταξιοδότηση. Χρειάζεται δουλειά και καμπάνιες ενημερώσεις για να συνειδητοποιήσουμε τη συνειδητοποιότητά μας. Το στίχημα είναι αν μπορούμε να μετατρέψουμε τη σχέση εργοδότη-εργαζομένου σε σχέση συνεργασίας μεταξύ μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνκα. Θα γίνει συζήτηση τώρα επί του σχεδίου έκθεσης της κυρίας Κούνεβα. Ποιος θέλει το λόγο. Η κυρία Λόπε Φοντανιά πρώτα. Σας ευχαριστώ. Αντικαθιστώ εδώ την κυρία Ρώσα Εσταράς, που δυστυχώς απουσιάζει και θα σας μεταφέρω τα δικά, τα δικά της σχόλια. Υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μορφών της οικιακής εργασίας, της αμοιβόμενης και μη. Η πρόσβαση των γυναικών στην εργασία μεταποδοχών εκτός της εστίας τους προκάλεσε την αύξηση των οικιακών εργασιών των αμοιβόμενων. Μία τέτοια γυναίκα μπορεί να καλύψει πολλές ανάγκες και απαιτήσεις. Βέβαια, περισσότερες δουλειές είναι μερικής απασχόλησης. Από αυτήν την άποψη και η μισθή των γυναικών αυτών ε, συνήθως ε, δηλώνονται ως έσοδα των γυναικών, δηλαδή προϋποθέτουν άλλες πηγές εσόδων. Επίσης θεωρούνται σχετικά ανειδίκευτες εργασίες. Δεν απαιτούνται ε, διπλώματα, πτυχία ή κατάρτιση. Ο καθένας ε, κάνει τη δουλειά του με βάση ε, τη, τα προσόντα του και το φύλλο του. Είναι ένας κλάδος που δεν έχει προσδιοριστεί επαρκώς. Πολλοί τέτοιοι απασχολούμενοι στις οικιακές εργασίες ε, υποτιμούνται. Υπάρχει σύγχυση μεταξύ του ιδιωτικού τομέα, στο οποίο γίνεται μια τέτοια δημόσια εργασία και μάλιστα ενό ξένου προσώπου που, που δεν προέρχεται από την ίδια την οικογένεια. Θα πρέπει να προβλεφθεί και ένα δημόσιο χώρο για την εργασία αυτή. Παρόλο που γίνεται σε ιδιωτικά σπίτια, θα πρέπει να αναγνωριστεί επίση ε, ο κλάδο αυτό τη οικιακή εργασία. Μόνο με τέτοια αναγνώριση θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε μεγαλύτερη δικαιοσύνη και στου μισθού και στι ε, εργασιακέ συνθήκε. Πρόκειται για μια εργασία που απαιτεί προσόντα. Παρόλο που μερικέ γυναίκε τη μόνη εμπειρία που έχουν είναι από τα δικά του σπίτια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει ρύθμιση αυτής της άτυπης ανεπίσημης μορφής εργασίας και να δούμε και τη μεταναστευτική πολιτική. Γιατί τέτοιε γυναίκε που κυρίω είναι μετανάστριε υφίστανται σε διακριτική μεταχείριση ό,τι αφορά τα εργασιακά του δικαιώματα. Εργάζονται με πολύ χαμηλού μισθού, που ε, ελάχιστα καλύπτουν ή πολύ περιορισμένα την κοινωνική ασφάλιση και πολύ συχνά οι εργαζόμενοι αυτοί αποκλείονται από τις προστατευτικά μέτρα ε, για τις απολύσεις συνήθως δεν ε, καλύπτονται από την εργασιακή νομοθεσία με ελάχιστες εξαιρέσεις σε κάποια κράτη-μέλη. Στις δυτικές χώρες και στις νότιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η οικιακή εργασία ρυθμίζεται περισσότερο με ειδικέ νομοθεσίες ή με συλλογικές διαπραγματεύσεις. Στην κεντρική Ευρώπη και στην ανατολική Ευρώπη έχουμε αντίθετα ε, ρύθμιση μέσω της εργασιακής νομοθεσίας. Αν κάνουμε ανάλυση των κανονισμών που ισχύουν και των νομοσχεδίων στις διάφορες χώρες για τα θέματα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχει μείωση της προστασίας σε ό,τι αφορά τις απολύσεις. Χρειαζόμαστε Υπάρχει επίσης μεγαλύτερη ελαστικότητα και ευελιξία και πολύ βραχυπρόθεσμε συμβάσει και τεράστια ευελιξία σε ό,τι αφορά τον μέγιστο αριθμό εργασιών ή τι απαιτήσει για τις υπερορίες ή τις, ε, ε, εκτός, ε, τις, τις μακρές μέρες, ώρες εργασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που είπατε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα ε, και θα ήθελα να πω και άλλα τρία πράγματα, αν μου επιτρέπετε, γιατί νομίζω ότι πρέπει να τα κουβεντιάσουμε. Το ένα είναι η βία, η βία που ασκείται έναντι αυτών των ατόμων. Γιατί, ξέρετε, επειδή ζουν όλοι μαζί στο σπίτι, αυτό συνεπάγεται και κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις για τις γυναίκες. Βεβαίως, ε, δεν είναι ότι κάθε φορά που μιλάμε για τις γυναίκες πρέπει να μιλάμε και για τη βία, αλλά σε αυτή την ε, ειδική περίπτωση πρέπει να μιλήσουμε για βία. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το θέμα ε, της αμοιβή. Πολλές φορές ε, στις γυναίκες αυτές του αφαιρούν το ότι τρώνε και ζουν στο σπίτι. Όμως αυτό δεν είναι σωστό. Τους παίρνουν τα μισά χρήματα γιατί απλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα δωμάτιο ή να φάνε με τους υπόλοιπους. Αυτό όπως σας είπα είναι άδικο. Και ενώ υποτίθεται ότι η αμοιβή είναι ικανοποιητική, τελικά οι γυναίκες παίρνουν τα μισά λεφτά. Το τρίτο που με ενδιαφέρει είναι η δομή, αν μπορείτε να μου πείτε, η ηλικιακή δομή εννοώ. Δηλαδή, από πλευράς ηλικία ε, οι γυναίκες ε, αυτές ε, σε ποιο ηλικιακό φάσμα εντάσσονται. Είναι νέες, είναι πολύ νέες οι γυναίκες αυτές. Δηλαδή, μήπως είναι τα κορίτσια εκείνα τα οποία πάνε να δουλέψουν και τελικά δεν μπορούν να σπουδάσουν. Αυτά είναι τρία θέματα που ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Ευχαριστώ. Η κυρία έχει το λόγο. Δεν περίμενα να μου ξαναδώσει το λόγο τόσο γρήγορα. Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να σας πω ότι η αντικαθιστώ τη συνάδελφο Τασούν, η οποία παρακολουθεί το θέμα και η οποία μου έχει γράψει κάποιες σημειώσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θέλω να πω το εξής. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς ε, που συζητείτε σήμερα το θέμα. Κυρία Κούνεβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που πολλές φορές το βάζουν κάτω από το χαλί και δεν το αποδίδουν τη σημασία που του προσήκει. Ε, λοιπόν πολλά και σημαντικά ερωτήματα. Το πρώτο για μας είναι αυτό που είπατε και εσείς κυρία Κούνεβα, δηλαδή το να σέβεται κανείς, να εκτιμά αυτή τη δουλειά. Γιατί η δουλειά αυτή παίζει καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική ένταξη. Η δουλειά αυτή γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Το να στηρίζει κανείς ανθρώπους είναι καθοριστική σημασία γιατί βλέπουμε ότι οι κοινωνίες μας διέρχονται μια δημοκρατική, δημογραφική, με δημογραφική αλλαγή. Πιστεύουμε λοιπόν ότι όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και ε, υπάρχει σαφώς μια θετική συμβολή στην κοινωνία και στην οικονομία από πλευράς αυτού του προσωπικού. Αυτό δεν φαίνεται όμως, δεν φαίνεται στην κοινωνία. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι κάτι ε, το οποίο έχει τη διάσταση του φύλου και πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Πάνω από το των ε, γυναικών σε οικιακές εργασίες είναι γυναίκες και κυρίως μετανάστριες. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι πολύ συχνά οι γυναίκες αυτές είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης, ε, είναι τροτές σε εκμετάλλευση η βία είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες μορφές εκμετάλλευσης και αυτό πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Και κάτι άλλο, όταν φτάνουμε στο ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε ή τι έχουμε να προτείνουμε για να αλλάξει η κατάσταση. Εδώ λοιπόν εμείς θα θέλαμε να υπάρχει εγγύηση για ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων, να υπάρχει κοινωνική ασφάλιση, κοινωνικές προδιαγραφές, προστασία από οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης, εγγύηση εγγυήσεις εχέγγυα στο οικιακό προσωπικό διότι επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά η εργασία του οικιακού προσωπικού είναι καθοριστική σημασία για την κοινωνία μας. Και κάτι το τελικό. Μέχρι τώρα μόνο τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυρώσει την σύμβαση του ILO, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για την οικιακή εργασία. Πρέπει λοιπόν να πιώσουμε όλα τα κράτη-μέλη να κυρώσουν αυτή τη σύμβαση, γιατί αυτό θα ήταν ένα πρώτο βήμα έτσι ώστε να μην υπάρχει εκμετάλλευση και δεύτερον να δείξουμε και να αναγνωρίσουμε ότι το οικιακό προσωπικό πραγματικά προσφέρει τα μάλα στις κοινωνίες μας. Αν θυγούν αυτά τα θέματα νομίζω ότι θα έχουμε προχωρήσει αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Κυρία Μπεσέρα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ζουμπέρ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κούνεβα για την έκθεσή της για ένα θέμα που μας αφορά όλους πιστεύω γιατί όλοι γνωρίζουμε κάποιον που απασχολείται σε αυτόν τον κλάδο τη οικιακή εργασία ή είναι προσωπικό φροντίδα. Όλε έχουμε βοηθού στο σπίτι, οικιακέ βοηθού ή που φροντίζουν κάποιον ε, οικείο μα. Γνωρίζουμε τι συνθήκε λοιπόν υπό τι οποίε εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ θα σα μεταφέρω τα σχόλια τη κυρία Λίνερ για αυτό το σχέδιο έκθεση. Πέραν το ότι πρόκειται για ένα θέμα πολυδιάστατο, γιατί το θέμα της οικιακή εργασίας ε, ε, είναι διαφορετικό από το θέμα των απασχολούμενων ε, σε τέτοιες δουλειές. Ε, πολλές γυναίκες, εκτός ότι είναι απασχολούμενες στην οικιακή εργασία και οι ίδιες έχουν, ασχολούνται με οικιακές εργασίες στο σπίτι τους. Είναι 80% αυτών των γυναικών. Και μιλούμε για εκατομμύρια γυναικών και κοριτσιών που απασχολούνται ως οικιακές βοηθοί σε ιδιωτικές κατοικίες και πέραν του σημαντικού έργου που διαδραματίζουν στην κοινωνία, για να μπορέσουν να συμμετέχουν στην αγορά εργασία, για να συνδυάσουν ε, τον προσωπικό με τον επαγγελματικό τους βίο, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε την πραγματικότητα ότι είναι η ομάδα που υφίσταται την περισσότερη εκμετάλλευση και τις περισσότερες καταχρήσεις και κακομεταχείριση. Και μάλιστα η σχετική σύμβαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασία μόνο από τέσσερι χώρε έχει εγκριθεί και έχει κυρωθεί. Γιατί οι υπόλοιπε 24 χώρε δεν κύρωσαν τη σχετική σύμβαση τη Παγκόσμια Οργάνωση Εργασία. Νομίζω χρειάζεται θέληση και αποφασιστικότητα και αυτό θα πρέπει να πετήσουμε από τα κράτη-μέλη. Να τηρηθούν οι υποχρεώσει, οι ανηλυμένε υποχρεώσει. Και τα κράτη-μέλη που ήδη έχουν έτοιμο το πακέτο αυτό ε, της σύμβασης ε, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας δεν έχουν παρά να την εφαρμόσουν. Επίσης θα πρέπει να, να αναγνωρίσουμε τον θετικό αντίκτυπο που, έχει σε, που έχουν σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο αυτή οι οικιακοί βοηθοί γιατί συμβάλλουν στην ε, ευεξία και στην ευημερία και την ατομική και την οικογενειακή και την κοινωνική. Ο απασχολούμενος στον κλάδο αυτό ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων φροντίζει το σπίτι, αλλά φροντίζει και ανθρώπους στο σπίτι. Βέβαια, άλλο η οικιακή εργασία και άλλο η φροντίδα παιδιών ή ηλικιωμένων ή ατόμων με κάποια εξάρτηση. Αυτό δεν είναι μια απλή δουλειά. Είναι ένα θέμα που επηρεάζει την ίδια την κοινωνία. Οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμίσουμε τον κλάδο αυτό. Είναι επιτακτική ανάγκη η ρύθμιση. Θα πρέπει να γίνει αμέσως. Επίσης θα πρέπει να καταπολεμήσουμε με συνεπή, συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο και τη σωματεμπορία και το εμπόριο ανθρώπων. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να προβλέψουμε ε, μια κατώτατη ηλικία, ένα ελάχιστο όριο ηλικία για τους απασχολούμενους στον κράτο αυτό, για να αποφεύγουμε ανήλικοι να απασχολούνται σε τέτοιες εργασίες. Αυτό δεν σημαίνει επίση ότι κάποιο που ασχολείται στον κλάδο αυτό θα πρέπει να στερείται άλλα στοιχειώδη δικαιώματα όπω είναι το δικαίωμα στην παιδεία για οποιαδήποτε γυναίκα ή οποιαδήποτε κορίτσι. Η κυρία Ροδρίγκε θα μα μιλήσει και για το σημείο αυτό αργότερα. Η παιδεία είναι κέριο ε, τομέα και παράγοντα για τη χειραφέτηση των γυναικών. Οπότε θα πρέπει να άρουμε τα εμπόδια και να φροντίσουμε διαφύλαξη αυτού του δικαιώματο στην παιδεία. Ένα άλλο σημείο σημαντικό, τις περισσότερες φορές οι εργασίες αυτές είναι αδήλωτες. Ανήκουν ε, στην ε, παραοικονομία πολλές φορές. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει και τους εργαζόμενους αλλά και την κοινωνία και το κράτος, ε, ο αδήλωτος χαρακτήρας αυτής της εργασίας. Επίσης θα πρέπει να ξεχνούμε τη σχέση που έχει ο κλάδος αυτός οικιακής εργασίας με τις εθνικές μεταναστευτικές πολιτικές. Γιατί ο περιοριστικός χαρακτήρας που επιβάλλουν πολλές χώρες για την οικιακή εργασία αφήνει πολλούς μετανάστες εγκλωβισμένους σε μια κατάσταση παράτυπης και αδήλωτης εργασίας. Σας ευχαριστούμε για την προθυμία σας να ακούσετε τις παρατηρήσεις μας και νομίζω ακριβώς ότι ο πολυδιάστατος χαρακτήρας αυτού του σημαντικού θέματος που έχει κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο ταυτόχρονα ε, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη και όλα αυτά τα σημεία θα συμβάλλουν στο να εμπλουτιστεί η έκθεση προκειμένου να αποκτήσει συνοχή και αρτιότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπεσέρα. Ακούσαμε πολλές παρατηρήσεις και σχόλια. Δεν βλέπω άλλον κανένα ζητάει το λόγο. Δεν ξέρω αν η συγκεκριά μας η κυρία Κούνεβα θέλει να σχολιάσει αυτά που άκουσε. ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Συμφωνώ με όλα όσα είπατε. Κάποιες απαντήσεις. Η βία είναι ένα φαινόμενο που πραγματικά υπάρχει και θα συνεχίζει να υπάρχει όσο τα δεν ρυθμίζεται το επάγγελμα αυτό. Αν καταφέρουμε να διασφαλίσουμε κοινέ αρχές, οι γυναίκες αυτές θα είναι δηλωμένες θα λαμβάνουν την αμοιβή τους χωρίς υποχρεώσει να μένουν μέσα στα σπίτια που εργάζονται και χωρίς υποχρεώσει διαπραγμάτευσης το μισθού τους. Γυναίκες όλων των ηλικιωμένων των όλων των δικαιωμάτων των ηλικιών, των ηλικιών συγγνώμη, απασχολούν, απασχολούνται στο κλάδο. Στόχος μας λοιπόν. λοιπόν να προστατεύσουμε όλες τις κατηγορίες. Αυτό για τώρα. Ευχαριστώ. Muito obrigada. Σας ευχαριστούμε κύριε Κούνεβα. Έγινε λοιπόν αυτή η ανταλλαγή απόψεων, πολύ χρήσιμη για να συγκεντρωθούν παρατηρήσεις που θα είναι χρήσιμες και για τη διαμόρφωση της έκθεσης. Η συζήτηση επί του σχεδίου έκθεσης θα γίνει στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2015 στην Επιτροπή μας. Περνάμε τώρα στο σημείο 5 της ημερήσης διάταξης. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες της έκθεσης με θέμα χειραφέτηση των γυναικών μέσω της παιδείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ψηφίσουμε αύριο. Θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Λιλιάνα Ροντρίγκε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ πορτογαλικά θα μιλήσω. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να διορθώσω τον τίτλο που έχει μεταφραστεί άσχημα στα πορτογαλικά. Καπασιτασάων δεν είναι ποντεραμέντου. Η χειραφέτηση δεν αποδόθηκε σωστά στα πορτογαλικά. γιατί ουσιαστικά περί πρόκειται και όχι απλώς απόκτηση κάποιων ικανοτήτων, αλλά πρόσβαση στην εξουσία ουσιαστικά. Το empowerment που λέμε στα αγγλικά. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους που συνέβαλαν με τις τροπολογίε τους. Ήταν θεμελιώδη σημασία η συνεισφορά τους προκειμένου να καταλήξουμε στις τροπολογίες στα στα σημεία αυτά. 206 τροπολογίες, 206 ιδέες δηλαδή που για, το, για την γνωμοδότηση αυτή. Η συμπίλησή τους οδήγησε σε 20 συμβαστικές τροπολογίες ε, και αυτές οι συμβαστικές τροπολογίες ήταν η μεγαλύτερη μας νίκη. Να θέσουμε στο επίκεντρο της συζήτησης το πιο σημαντικό. Τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες και το ρόλο της παιδείας στη χειραφέτησή τους. Και μάλιστα έχουμε και τη Διεθνή ημέρα της γυναίκας ε, που έθεσε ως προτεραιότητα την παιδεία που είναι σημαντικό στοιχείο ελευθερίας και χειραφέτησης. Γιατί η παιδεία βέβαια δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά είναι ένα μέσο που επιτρέπει την εξασφάλιση της αυτονομίας και της ελευθερίας που δεν διδάσκεται αλλά αποκτάται. Επίσης είναι ένας μακρύς δρόμος που γίνεται με την παιδεία την και την κατάρτιση. Δεν μπορούμε να ξεκινάμε προθύστερα σχήματα θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα εφόδια που δίνει η παιδεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι αυτά που είναι στην καλύτερη θέση να εξασφαλίσουν μια δημοκρατική πρόσβαση στην παιδεία. Εκπαιδεία και εκπαίδευση για την αυτονομία και την ελευθερία. Βέβαια πολλές φορές έχουμε σχολικές κουλτούρες που δεν θεωρούν την ελευθερία ως πρωταρχική αξία. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε αυτά τα στοιχεία υπόψη την παιδεία και την δικαιοσύνη που θα πρέπει να ισχύει. Επίσης, μας ανησυχεί το γεγονός ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες ακόμη υφίστανται διακριτική μεταχείριση σε μια Ευρώπη που υποτίθεται είναι πολιτισμένη και έχει θεμελιώδεις αρχές και αξίες και παρόλα αυτά δεν έχει ολοκληρώσει αυτό το, το τρίπτυχο της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης. Δύο είναι οι βασικοί στόχοι τη ε, γνωμοδότηση. Να εξασφαλίσουμε μέσω τη παιδεία τη χειραφέτηση των κοριτσιών και των γυναικών, να τηρήσουμε τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη που θεωρεί την παιδεία ω βασικό εφόδιο για την ε, αποφυγή τη της ε, διάκρισης μεταξύ των δύο φύλων και θέλουμε μια σχολική κουλτούρα ισότητας των φύλων, έλεγχος του εκπαιδευτικού προγράμματος προκειμένου να διευκολυνθεί καλύτερη λήψη των ε, επαγγελματικών αποφάσεων, να βελτιωθεί πρόσβαση των γυναικών ε, σε σημαντικές ηγετικές ε, θέσεις και να προωθηθεί η ισότητα και η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών. Επίσης, θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα μέτρα για να υλοποιηθούν οι προσανατολισμοί του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η πρόθεση των ε, μαθημάτων ε, των θετικών επιστημών ε, μηχανικής και άλλα να αποφευθούν τα στερεότυπα στα προγράμματα σπουδών, να έχουμε και στην κατάρτιση των καθηγητών το θέμα της ισότητας των φύλων, πρόθεση εγχειριδίων που θα εξασφαλίσουν αυτήν την ισότητα των ευκαιριών, πρόθεση κουλτούρας σχολικής που θα σέβεται την ισότητα των δύο φύλων, επίσης διαπαιδαγώγηση και των γονέων στην ισότητα των φύλων, βελτίωση του ποστού των γυναικών ε, ε, στις, δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οικονομική αρρωγή των οικογενειών προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των κοριτσιών στα σχολεία. Βέβαια, είναι φυσιολογικέ μερικέ φορέ οι διαφορέ και η διάσταση απόψε μεταξύ μα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε όλε οι κοινοβουλευτικέ δυνάμει και γι' αυτό χαίρομαι για τι 20 συμβαστικέ τροπολογίε τι οποίε καταφέραμε να καταλήξουμε. Ε, γιατί όλοι είμαστε υπέρ της λήψης συγκεκριμένων μέτρων για την κατάρτιση, για παράδειγμα, όλων όσων έμεσα ή άμεσα συμμετέχουν στην εκπαιδευτική κοινότητα. Από το πρόγραμμα σπουδών, επίσημο ή άτυπο, αλλά και του άδειλου προγράμματος, ε, που θα πρέπει και αυτό να συμβάλλει στη χειραφέτηση. Επίσης, ίση πρόσβαση στις πληροφορίες, στις ε, τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίες Και ανάπτυξη του πνεύματος ε, του ηγετικού πνεύματος και στις γυναίκες. Θα πρέπει στα προγράμματα αυτά ισότητας των φύλων να, ενισχυθεί ε, η διάσταση των δύο φύλων και η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το θέμα του προγράμματος που εδώ είναι πολύ σημαντικό γιατί εκεί ε, έχουμε το σχετισμό των δυνάμεων. Γι' αυτό και είμαι υπέρ της αλλαγής του τίτλου στην πορτογαλική μετάφραση, ώστε να λέμε χειραφέτηση και empowerment δεν θα πρέπει να έχουμε διάκριση μεταξύ ε, αρχηγών και υποτελών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ισότητα μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών. Γιατί χωρίς τη συμμετοχή των κοριτσιών δεν θα έχουμε πραγμάτως της ιδέας της ισότητας. Είναι σημαντικό σε μια τέτοια γνωμοδότηση να συμπεριλάβουμε και τους άνδρες. Γιατί χωρίς τη συμμετοχή τους δεν θα μπορούμε να μιλούμε για ισότητα των δύο φύλων. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, τη συμβολή σας ε, στη γνωμοδότηση αλλά και στο μέλλον της Ευρώπης. Η γνωμοδότηση αυτή δεν είναι δικιά μου, δεν είναι του σοσιαλιστών και δημοκρατών. Δεν στηρίζεται στην ε, διάσταση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Είναι μια κοινή γνωμοδότηση γιατί ε, είναι η έκθεση όλων όσων θέλουν, θεωρούν επιτακτική ανάγκη να συμβάλλουν στη χειραφέτηση των γυναικών με τους παιδείας, για να μπορέσουν τα κορίτσια να γίνουν χειραφετημένες γυναίκες. Θέλουμε να προστατεύσουμε τα κορίτσια, τις κόρες της Ευρώπης. Μ' αρέσει πολύ αυτή η έκφραση. Επίσης, ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις και ελπίζω αύριο να υπερψηφιστεί η έκθεση. Γιατί το δικαίωμα στην παιδεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι δικαίωμα των γυναικών, των κοριτσιών και όλων των παιδιών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ροντρίγκε. Τα σχόλιά σας για την πορτογαλική μετάφραση του, της γνωμοδότησης σημειώθηκαν, καταγράφηκαν από τη γραμματεία και θα ληφθούν υπόψη και να περάσουμε στη συζήτηση. Το λόγο έχει η κυρία Γκάλ Πέλτς. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά ε, την συγκητρία για αυτή τη συνεργασία η οποία ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική και θέλω να σας πω ότι πετύχαμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα και το έγγραφο αυτό ε, εκφράζει ακριβώς αυτά τα αποτελέσματα. Ε, θέλω να επισημάνω ότι ο στόχος όλων μας είναι ε, να υπάρχει υψηλό επίπεδο παιδείας και πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα και στις γυναίκες και στους άντρες να έχουν πρόσβαση στην παιδεία και η πρόσβαση αυτή είναι σημαντική όχι μόνο γιατί με τον τρόπο αυτό οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη ευκολία να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους αλλά και διότι ε, με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της φτώχειας. Η παιδεία και η πρόσβαση στην παιδεία είναι κινητήρια δύναμη της οικονομίας και κατόπιν τούτου η παιδεία η εκπαίδευση των γυναικών έχει πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζουμε, νομίζω ότι σε αυτό το τομέα μπορούμε να επενδύσουμε και να περιμένουμε αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε μια κοινή γραμμή και μπορούμε να εκπέμψουμε ένα κοινό μήνυμα έτσι ώστε να επιτευχθεί πρόοδος. Ε, η ισότητα των δύο φύλων είναι πολύ σημαντική, όπως και οι δείκτες, γιατί χρειαζόμαστε μελέτες που να καταδεικνύουν ε, την αποτελεσματικότητα όλων αυτών των μέτρων. Είναι εξάλλου σημαντικό ε, να είναι κατανοητό ότι και οι πόροι είναι καθοριστικής σημασίας. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να διατεθούν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία και εμείς ε, καλούμεθα να τα ε, αξιολογήσουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά. Αυτά είχα να πω και να επισημάνω για μια φορά ότι το έγγραφο είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Σας ευχαριστούμε κυρία Δεσέρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να ασχολούμαστε με τόσο πολυδιάστατες εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις, γιατί μας δίνουν ευκαιρία στενής και καρποφόρα συνεργασίας, όπως έγινε με τη γνωμοδότηση της κυρίας Ροντρίγες. Όσο πιο πολύμορφη και πολυδιάστατη είναι μια έκθεση και όσο περισσότερες ε, τροπολογίες κατατίθενται, τόσο περισσότερες ευκαιρίες υπάρχουν για να την εμπλουτίσουμε. Ήταν ε, υποδειγματική η διαδικασία των ε, τροπολογιών επ' ευκαιρία αυτής της έκθεσης. Και στην ημέρα, το Παγκόσμια ημέρα των γυναικών είχαμε και σεμινάριο, είχαμε ακρόαση και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι σημαντικό να εμπλέκουμε εδώ όλους τους ενδιαφερόμενους. Γιατί η γνωμοδότηση πέραν ότι ασχολείται με πολύ κρίσιμα ζητήματα, περιέχει και ένα βασικό μήνυμα, το ότι η παιδεία είναι το σημαντικότερο, το θεμελιώδες, ο θεμελιώδης παράγοντας για την αυτονομία και την ανεξαρτησία. Χωρίς πρόσβαση δεν εννοείται ούτε αυτονομία ούτε ανεξαρτησία. Γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πρόσβαση, ίση πρόσβαση όλων των κορισιών και των γυναικών στην παιδεία. Επίσης το περιεχόμενο της ε, παιδείας αυτής θα πρέπει να είναι κατάλληλο γιατί προστεί η πρόσβαση ε, σε μια παιδεία που το περιεχόμενό της θα είναι κατάλληλο. Δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την καρποφόρα διαδικασία που, ε, κατά τη συζήτηση της έκθεσης και τη σύγκληση που επιτεύχθη και επίσης ε, να εξάρουμε αυτή τη σημασία, τη σημασία που έχει η παιδεία για την αυτονομία και την ανεξαρτησία. Γι' αυτό και θα πρέπει σε όλα τα προγράμματα σπουδών να περιλάβουμε και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τη διαπαιδαγώγηση για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Οι γυναίκες, τα κορίτσια θα πρέπει να γνωρίζουν το σώμα τους και να έχουν τον έλεγχο του σώματός τους. Όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Από τη στιγμή που τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, θα γνωρίζουν ε, το σώμα τους, ε, σε τι χρησιμεύει, πώς μπορούν να, ε, να ζουν με αυτό, τι αλλαγές θα παρατηρήσουν και πόσο σημαντικές είναι αυτές οι αλλαγές στη ζωή, γιατί το σώμα το έχουμε για όλη μας τη ζωή. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία του. Αν όλα αυτά τα σημεία δεν, υπάρχουν, δεν βρουν τη θέση του στο πρόγραμμα σπουδών, πώς θα μπορούμε να μιλούμε για μια εκπαίδευση που θα βοηθά τις γυναίκες να χειραφετηθούν και να αποκτούν αυτή την εξουσία, το empowerment που λέμε στα γαλλικά. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι η κατάργηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων και στα σχολεία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, προ, προβάλλουν μοντέλα και επίσης κατάργηση των στερεοτύπων και στη διαφήμιση. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ισότητα των δύο φύλων μεταξύ των εκπαιδευτών. Γιατί πώς μπορούμε να προβάλλουμε ένα μοντέλο ισότητα στην κοινωνία αν ε, δεν έχουμε κάνει την προεργασία και σε επίπεδο εκπαιδευτών διδακτικού προσωπικού. Η παιδεία είναι το πιο σημαντικό από όλα και χρειαζόμαστε μια ολιστική σφαιρική προσέγγιση. Δεν είναι ε, μόδα η λέξη ολιστικός, σφαιρικός, αλλά σε όλους τους τομείς χρειάζεται και πάνω απ' όλα στην παιδεία αυτή η σφαιρική προσέγγιση. Η κυρία Μάλιγκαρκ από την QNGL. Eh, Ευχαριστώ. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Για μια έκθεση επί της οποίας εργαστήκαμε από κοινού με πολύ επικατομητικό τρόπο και καταλήξαμε και σε πολλές συμβαστικές τροπολογίες και σας ευχαριστώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα μα, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι εξαιρετικά σημαντικό για να ενισχύσουμε τι εργασίε μα σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο μιας πατριαρχικής ε, κοινωνίας βλέπουμε ότι οι άντρες κατέχουν την εξουσία εδώ και αιώνες. Και είναι θεμελιώδη σημασία να αλλάξει αυτός ο συσχετισμός δύναμης μεταξύ των φίλων. Και μέσω της εκπαίδευσης μπορούμε να διασφαλίσουμε αυτή την αλλαγή. Και έτσι θα έρθει και η ανεξαρτησία, η χειραφέτηση. Πρέπει να δώσουμε τέλος στα στερεότυπα, να δώσουμε 100 δυνατότητες να αναπτύξουν τις δυνατότητες τους τα παιδιά και όχι μόνο δύο. Ευχαριστώ λοιπόν την εισηγήτρια για τα όσα έχει κάνει. Και να επισημάνω ορισμένα στοιχεία στα οποία τελικά δεν ε, συμφωνήσαμε. Για παράδειγμα, μια τροπολογία που εμείς έχουμε προετοιμάσει, την 132, για τα μαθήματα φεμινιστικής αυτοπροστασίας. Είναι ένα νέο κόνσεπτ, μια νέα ιδέα, αλλά είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι ένα μέσο που θα μας ε, επιτρέψει να προετοιμαστούμε απέναντι στη βία. Είναι σημαντικό στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, λοιπόν, να υπάρχει και αυτό το μάθημα της αυτοάμυνας των γυναικών, γιατί έτσι θα εκπαιδεύσουμε τις νέες γυναίκες, τα κορίτσια, ε, να μάθουν να ψητεύουν τον εαυτό του και έτσι να διασφαλίσουν και τη θέση του στην κοινωνία. Αυτό δεν αφορά το σώμα, αλλά όχι μόνο το σώμα. Αφορά και την παρενόχληση. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντική αυτή την ιδέα και συνδέεται με αυτή την δυνατότητα δράση. Τροπολογία 132 λοιπόν. Ίσως δεν το γνωρίζετε, αλλά στη Σουηδία και στη Χιλή είναι από τις χώρες ε, με πλέον ιδιωτικοποιημένο εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μου. Έχουμε λοιπόν αυτό τον κίνδυνο τώρα τα σχολεία μας να γίνουν εταιρείε ουσιαστικά ε, εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο κίνδυνος. Σήμερα τα χρήματα του φορολογουμένου πηγαίνουν βέβαια στα σχολεία, αλλά τελικά καταλήγουν στις τσέπες των μετόχων. Είναι τρομερό αυτό το πρόβλημα και αυτό αναφέρεται και στην ε, τροπολογία 112 όπου επιμένουμε ότι τα δημόσια κονδύλια δεν πρέπει να καταλήγουν στις τσέπες των μετόχων. Σουηδία και Χιλή λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι οι χώρες ε, με τα πλέον ε, ιδιωτικοποιημένα εκπαιδευτικά συστήματα. Μετά, στην 146 τροπολογία αναφέρομαι στην ε, θετική προβολή των, ε, της ομάδας LGBT. Γιατί βλέπουμε ότι η ομοφοβία αυξάνεται και τα νέα αυτά άτομα πολλές φορές έρχονται αντιμέτωπα, αντιμέτωπα, αντιμέτωπα με αρετσιστικές ε, αντιδράσεις αυτό αφορά και τους ε, ομοφιλόφιλους και τους διεμφυλικούς, όλα τα αυτής κατηγορίας και πρέπει να προβάλλεται μια θετική εικόνα αυτής της ομάδας, αυτής της κατηγορίας πολιτών. Αυτό και στο πλαίσιο της φεμινιστικής μας θέασης. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πληρέστατη αυτή έκθεση ε, που θα ψηφιστεί και στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια, ελπίζω. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των Πρασίνων, η κυρία Χένκ. Ευχαριστώ. Πολλά και σημαντικά έχουν ήδη ακουστεί. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Να τονίσω μόνο κάτι το οποίο ανέφερε και η κυρία Μπιόρκ. Είναι πολύ σημαντικό για μας να συμπεριλάβουμε ιδίως στην κατάσταση ε, των νέων LGBT. Και πάλι παραμένουν ανησυχητικά υψηλά τα ποσοστά αυτοκτονιών στο πλαίσιο αυτής της ομάδας, ιδίως σε ό,τι αφορά ε, τους νέους ε, transsexual, που πραγματικά δέχονται τεράστιες πιέσεις ε, και στα σχολεία τους και πρέπει να προστατεύσουμε αυτά τα μέλη αυτής της κοινότητας και να πετύχουμε τους ε, στόχους που αναφέρονται στην έκθεση. Πρέπει λοιπόν στο σχολικό πρόγραμμα να ε, διδάσκεται και ο σεξουαλικός προσανατολισμός, Και είναι πολύ σημαντική η συμπερίληψη αυτού του στοιχείου στην έκθεση, γιατί υπάρχει πολύ σημαντικό ζήτημα με αυτό το θέμα σε σχολεία που υπάρχουν υψηλέ διακρίσει, μεγάλε διακρίσει μάλλον κατά αυτών των ατόμων και θα πρέπει να εύσουσουμε τη φωνή μας για να προστατεύσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις διακρίσει κατά αυτών των ατόμων. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κόμπερν από το EFTD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση θέλει περισσότερη γραφειοκρατία ουσιαστικά, περισσότερους φραγμούς ε, στα, ε, στο εκδοτικό σύστημα, ενώ η διδασκαλία θα πρέπει να είναι ο δικός μας στόχος και καλή μάλιστα και για ένα ετήσιο βραβείο για την ισότητα μεταξύ των φίλων. Σίγουρα όλοι εκείνοι που εξαρτώνται από τις ε, επιστηστικές τράπεζες για να επιζήσουν, σίγουρα θα μας συγχαρούν για τις επιλογές μας. Βλέπουμε ότι η στάση των μαθητών μπορεί πολλές φορές ε, να αποβεί σε βάρος τους. Τελικά θα κάνουμε, θα ε, κατηγορήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τους μαθητές. Μετά στην τροπολογία 39 λέμε ότι πρέπει να υπάρχει πολύ πιο στενή συνεργασία και να υπάρξει ανακατανομή της φροντίδα στην οικογένεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρέμβει στη, στον ιδιωτικό βίο ε, γάμων, ζευγαριών και οικογενειών. Μετά, θέλουμε αναφέρει κάποια τροπολογία, συγκεκριμένες ε, εκστρατείες ενημέρωσης και στα σχολεία για τους ε, αντίστοιχους ρόλους αγοριών και κοριτσιών στην οικογένεια. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να πείτε στα παιδιά πότε πρέπει να ξεκινήσουν ε, την οικογένειά τους και πώς να ζήσουν τη ζωή τους. Τροπολογία 132 προτείνεται η εισαγωγή των μαθημάτων αυτοάμυνας ε, των γυναικών. Τι ακριβώς σημαίνει αυτοάμυνα, φεμινιστική αυτοάμυνα. Βεβαίως να μάθουν οι νέοι πειθαρχία, αλλά η πολιτική προπαγάνδα τι σχέση έχει εδώ. Πραγματικά δεν έχει καμία απολύτω σχέση. Και τέλος, τροπολογία 141, 143 και 161 θέλουν σεξουαλική εκπαίδευση στο σχολείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίε και κύριοι, δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρέμβει στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών. Ευτυχώς δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε μεταφορικά, ούτε κυριολεκτικά, ε, να ε, επιβάλλει εκπαιδευτική πολιτική. Ελπίζω πραγματικά να μην υιοθετηθεί ούτε αυτή η έκθεση, ούτε αυτέ οι τρελέ τροπολογίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συγχωρώ, Πέτυρ του ΠΠΕ. Η κυρία Πετήρ από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με όσους είπαν ότι είναι κακή η μετάφραση σε μερικές γλώσσες, το ίδιο και στα κροατικά. Θα πρέπει να διορθωθεί η μετάφραση, να φροντίσουμε να είναι πιο ποιοτικές οι μεταφράσεις για να καταλαβαίνουμε και για τι πράγμα μιλάμε. Επίσης θα ήθελα να πω ότι είναι σαφής η πρόθεση της εισηγήτριας που θέλει να συμβάλλει στη χειραφέτηση των γυναικών, των κοριτσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της παιδείας. Βέβαια είναι κάπως ολισθηρό το έδαφος αυτό. Θα πρέπει να φροντίσουμε, ναι, να βελτιώσουμε τη θέση των κοριτσιών και την πρόσβασή τους στην παιδεία, αλλά να μην ε, παρέμβουμε στις ε, αποκλειστικές αρμοδιότητες των κρατών μελών, γιατί θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επικουρικότητα και η παιδεία και η οικογένεια είναι θέματα που επαφίονται στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα επίσης να προτείνω στην εισηγητριά και κατέθεσα και σχετικές τροπολογίες, ε, γιατί είναι σημαντικό να εκεί που μιλούμε για την παιδεία των κοριτσιών, να στηριχθούμε σε πολύ σημαντικές συμβάσεις, ε, πολύ σημαντικές συμβάσεις για τα κορίτσια. Και στη δική μου τροπολογία αναφέρω τη μνήα στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Και θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε στο προήμιο, στις αιτιολογικές σκέψεις, εκτός της μνήας ε, της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Παιδιών, να μιλήσουμε και για την ε, διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την Διεθνή Σύμβαση για τα πολιτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα του πολίτη. Επίσης και το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε και τα έγγραφα αυτά στην σημαντική γνωμοδότηση, να παραπέμπουμε σε αυτά και να φροντίζουμε να τηρούνται όλες αυτές οι συμβάσεις, ιδιαίτερα όταν μιλούμε για το δικαίωμα των κοριτσιών στην παιδεία. Κατά τη γνώμη μου, η γνωμοδότηση ε, παραλείπει κάτι που είναι πολύ σημαντικό, σημαντικό και για μένα αλλά και για όλους τους ε, συμπολίτες μου. Ε, τα, οι έχουν δικαίωμα και ευθύνη για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Κάτι που αναφέρει και το άρθρο 18 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Και γι' αυτό κατέθεσα τροπολογία, τη τροπολογία υπαριθμών 76, γιατί ίσως ακούσει χωρίς να το θέλετε, παραλείψατε το δικαίωμα των γονιών και την ευθύνη των γονιών για την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους και την, ε, τον έλεγχο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Γιατί οι γονεί ε, και οι κυδεμόνε των παιδιών είναι αυτοί που κατά πρώτο λόγο έχουν την ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών και την διαπαιδαγώγησή τους. Και αυτοί φροντίζουν πρώτα για την ευημερία των παιδιών τους. Γι' αυτό σας παρακαλώ να δεχτείτε την τροπολογία μου υπαριθμών 76 και να τη συμπεριλάβετε στην αγνωμοδότησή σας, γιατί επαναλαμβάνω κατοχυρώνεται από σημαντική σύμβαση που σας προανέφερα. Γιατί τα πιο σημαντικά πράγματα τα μαθαίνουμε στην οικογένεια, στο σπίτι, από τους γονείς. Εκεί μαθαίνουμε τι άνθρωποι θα γίνουμε. Και αργότερα το σχολείο βοηθάει και συμπληρώνει αυτή τη διαπαιδαγώγηση. Αλλά ξεκινάει από τους γονείς, από το σπίτι, από την οικογένεια. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ζυπνάνσκα. Eh, θα ήθελα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και όλους τους ε, άλλους σκιώδης ηγητές. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι μας θέλουμε να υπάρχει ισότητα ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες και η παιδεία είναι αναμφίβολα ένας τρόπος για να επιτύχουμε την ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες και επίσης και η παιδεία μπορεί να οδηγήσει στην καταπολέμηση της φτώχειας. Θα ήθελα εξάλλου να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω θερμά για τις τροπολογίες που καταθέσατε και όπου γίνεται λόγος για τα κορίτσια τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στην ε, παιδεία. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστώ θερμά και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κυρίως ε, τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνουμε στι αρμοδιότητε των κρατών μελών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η παιδεία εξακολουθεί να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Άρα δηλαδή το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προβαίνουμε σε συστάσει. Είναι αλήθεια ότι οι γονείς είναι κυρίως υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των παιδιών και γι' αυτό ε, οι τροπολογίες 76 και 78 όπου γίνεται λόγος για το βασικό δικαίωμα των γονέων να επιλέγουν εκείνη την εκπαίδευση των παιδιών τους ε, έτσι ώστε ε, να μην ε, αποδίδεται το σύνολο των αρμοδίτων για την εκπαίδευση στα σχολεία. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι η οικογένεια θα πρέπει να είναι η βάση της ε, παιδείας. Εγώ προσωπικά είμαι μητέρα, έχω τρία παιδιά και γνωρίζω ότι η ανατροφή στο σπίτι είναι καθοριστική σημασίας. Το να συμπεριλαμβάνονται και τα αγόρια στις οικιακές εργασίες και να εκπαιδεύονται για τις ε, σχέσεις τους ε, με τις ε, γυναίκες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζήτησε το λόγο για να δευτερολογήσει η κυρία Μπεσέρα, αλλά τη θέμα παρακαλώ να είναι λακωνική. Μία σύντομη παρατήρηση θα ήθελα να κάνω, μία απάντηση στον κύριο Κοβούνη και στην κυρία Πετήρ. Η διαφορά μεταξύ της διαδικασίας που ακολουθεί και στην έκθεση και της στιγμής Τη σημερινή είναι ότι ήδη έχουμε εγκρίνει τη στρατηγική 2016-17 20 για την ισότητα. Αυτό είναι το πλαίσιο, αυτή η στρατηγική ε, μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε τη στρατηγική μας θέση και τι εμπίπτει στις κοινοτικέ αρμοδιότητες και τι όχι. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με την επικουρικότητα. Στο πλαίσιο αυτών των στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών που έχουμε και που εγκρίναμε, Αυτές τις κατευθυντήρες γραμμές θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Αυτά είναι τα σημεία αναφορά μας για να, να ξέρουμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε και τι είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι όχι. Ευχαριστώ. Κύριε Κόμπορτ, αλλά παρακαλώ επιγραμματικά, γιατί δεν μας έχει μείνει πολύ χρόνο. Κύριε Πρόεδρε, σας υπόσχομαι ότι θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ε, θέλω να σας πω ότι δεν είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να παρεμβαίνουν στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών. Όταν η Μεγάλη ήρθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπήκε όχι για να λέει στου ανθρώπου πώ να ζουν τη ζωή τους, τι να κάνουν με τα παιδιά τους ε, ή αν θέλετε για να επικρίνει τα εκπαιδευτικά του συστήματα. Αυτό είναι κάτι που αφορά μόνο τα κράτη-μέλη. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι η εκπαίδευση δηλαδή, που αφορά το Κοινοβούλιο καμία σχέση. Μάλιστα. Θα ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Thank you. Um, Angelos Agalianos from DG Education and Culture. Um, This ε, κοιτάξτε, είναι μια πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε να σημειώνεται πρόοδο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι μια δουλειά η οποία εντοπίζει πάρα πολλά βασικά θέματα και λύσεις. Ε, όλο αυτό δείχνει ότι η ισότητα των δύο φύλων δεν προκύπτει από μόνη της, δεν είναι τυχαία Βλέπουμε λοιπόν ότι παραμένουν προκλήσεις στα ευρωπαϊκά εκποτεκτικά συστήματα για την ισότητα των δύο φυλών και βλέπουμε και μία άλλη διάσταση που είναι η χρήση της ε, εκπαίδευσης ως ένα θεμελιώδες εργαλείο για την κοινωνική αλλαγή στις κοινωνίες μας. Επίσης βλέπουμε το ρόλο της εκπαίδευσης για τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που μας συμπεριλάβατε μέχρι τώρα σε όλες τις φάσεις. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτό. Περιμένουμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα και τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν σε συγκεκριμένες πολιτικές. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε πολλά σχόλια, πολλές παρατηρήσεις. Δεν ξέρω αν η συγκεκριά μας θέλει πάλι το λόγο. Βέβαια δεν έχω χρόνο για να απαντήσω διεξοδικά και μεμονωμένα σε όλες τις παρατηρήσεις. Νομίζω ότι το σημαντικότερο ήταν ο ήρεμος και νυφάλιος διάλογος που είχαμε μεταξύ μας καθ' όλη τη διάρκεια των διαβουλεύσεων. Με πολύ πολιτισμένο, νυφάλιο και ψύχρεμο τρόπο κάναμε τις συζητήσεις και καταλήξαμε στο σημερινό τελικό αποτέλεσμα. Βέβαια, η γνωμοδότηση αυτή σε καμία περίπτωση θέλει να παρέμβει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, ούτε να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν οτιδήποτε μέτρο. Προβαίνει σε συστάσεις απλώς η γνωμοδότηση. Αυτό θα πρέπει ε, να τονιστεί. Εμείς ε, συστήνουμε το κατάλληλο, κατά τη γνώμη μας, για τα κορίτσια και τα αγόρια σε ό,τι αφορά την ε, παιδεία. Θα μπορούσαμε βέβαια να συνεχίσουμε τις ε, συζητήσεις για να τελειοποιήσουμε ακόμη περισσότερο την έκθεση. Αλλά νομίζω ότι η τελική εκδοχή καλύπτει σε μεγάλο βαθμό όλους όσους κατέθεσαν ε, τροπολογίες από όλα τα πολιτικά κόμματα. Κύριε Μπερκ, δεν έχουμε αφαιρέσει το θέμα των μαθημάτων αυτοάμυνας το έχουμε σε παρέθεση, ίσως το βελτιώσουμε, αλλά προβλέπεται γιατί θεωρούμε σημαντικό να αναπτυχθούν όλα τα εφόδια και όλα τα, όλες οι ικανότητες των κορισιών και οι σωματικές. Γι' αυτό και αναφέρθηκε το θέμα της αυτοάμυνας, αλλά και το θέμα των ΛΟΑΔΜ. Και αυτό συζητήσαμε στις συμβαστικές τροπολογίες. Αν θα πρέπει να έχουμε ένα κατάλογο, αλλά ήταν ανησυχητικό να με μερικούς κατά μέρο. Γιατί ήταν σαφείς οι διαφορές που υπήρχαν σε όλη την έκθεση. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν με τις τροπολογίες τους στη διαμόρφωση της έκθεσης και ελπίζω αύριο να καταφέρουμε να υπερψηφίσουμε την, την γνωμοδότησή μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η ψηφοφορία της έκθεσης αυτής θα λάβει χώρα αύριο στις 10. Περνάμε στο σημείο 6 τώρα και θα ήθελα να ζητήσω από τους καλεσμένους μας να έρθουν στο Προεδρείο και να λάβουν θέση. Το σημείο 6 λοιπόν προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με θέμα τις νέες κατευθυντήρες γραμμές και τη συμπερίληψη στην ανθρωπιστική δράση, τις παρεμβάσεις ε, για την καταπολέμηση της βίας ε, ε, εις βάρος του άλλου φίλου. Στις 31 Μαρτίου αποφασίσαμε στην Επιτροπή να οργανώσουμε ανταλλαγή απόψεων με τη UNICEF για να μας παρουσιάσει τους νέους προσανατολισμούς, τις νέες κατευθυντήρες γραμμές, για να περιλάβουμε στην ανθρωπιστική μας δράση τις ε, παρεμβάσεις μας ε, και τις ενέργειες μας για να αποφευθεί η βία μεταξύ των δύο φύλων. Καλέσαμε μάλιστα τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, την πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, την κυρία Λίντα Μάκαβαν, για να συμπροεδρεύσει, αλλά Δυστυχώς ε, δεν ε, μπόρεσε να έρθει η κυρία Μάκαβαν. Μας έστειλε όμως τον αντιπρόεδρο ε, το, της Επιτροπής Ανάπτυξης, τον κύριο Κούλογλου, ο οποίος βρίσκεται στα αριστερά μου. Θεωρούμε ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα συμβάλλει στην διαμόρφωση της γνωμοδότησης που καλούμαστε να συντάξουμε στην έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης για την προετοιμασία της ε, Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής ε, με θέμα της προκλήσης ε, της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Βοήθειας και τη γνωμοδότησή μας θα τη συντάξει η κυρία Χέντ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Έχουμε καλέσει εκπροσώπους οργανώσεων και θα δώσω πρώτα το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ αγαπητοί Ινές, αγαπητοί συνάδελφοι και καλεσμένοι. Εκ μέρους της ε, Επιτροπής Ανάπτυξης σας καλωσορίζω. Πιστεύουμε ότι αυτές οι νέες οδηγίες ε, που παρουσιάζονται στο Κοινοβούλιο είναι πολύ επίκαιρες τα νέα και οι εκθέσεις που έχουμε από ανθρώπους ε, που δουλεύουν στα διάφορα σημεία συγκρούσεων μας δίνουν εικόνες και ιστορίες μεγάλης ανθρώπινης τραγωδίας από συγκρούσεις που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι άνθρωποι. Όπως έχουμε δει στην δημοκρατία του Κονγκό και στο Σουδάν και τώρα βλέπουμε στο Ιράκ και τη Συρία είναι οι πιο ασθενείς κατηγορίες του πληθυσμού, δηλαδή οι γυναίκες και τα κορίτσια που βαστάνε το μεγαλύτερο βάρος των πολέμων και των συγκρούσεων απαγωγές, σεξουαλική εκμετάλλευση, βιασμοί, σκλαβιά, κυκλοφορία γυναικών και αναγκαστική γάμη είναι ορισμένα από τα πράγματα που μαθαίνουμε και κάνουν εξαιρετικά επίκαιρη την ανάγκη να υπάρξει προστασία των γυναικών και των κοριτσιών αυτές όλες οι συγκρούσεις που παρακολουθούμε δεν είναι ουδέτερες. Έχουν διαφορετική συνέπεια ανάλογα με το αν τα θύματα είναι άντρες, γυναίκες, νέοι ή κορίτσια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να δούμε ειδικά και να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε να προστατεύσουμε αυτά τα πολύ ευαίσθητα και ευάλωτα θύματα των συγκρούσεων. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτές οι οδηγίες θα αποτελέσουν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα πλαίσια της συνολικότερης προσπάθειας αντιμετώπισης των ανθρωπιστικών ε, κρίσεων. Σας ευχαριστώ πολύ και δίνω στην ΕΝΕΣ το... την Προεδρία. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους καλεσμένους μας και εκ μέρους Επιτροπής των Γυναικών να σας ε, ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας για τη συμμετοχή τους στη συζήτηση. Να δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Γκουίν Λιουίς από το πρόγραμμα της UNICEF για 10 λεπτά παρακαλώ. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Έχω προετοιμάσει για ένα PowerPoint. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε εδώ σήμερα. Αυτές οι κατευθυντικές γραμμές είναι εξαιρετικά σημαντικές για εμάς και θεμελιώδη σημασία για τη UNICEF. Χαιρόμαστε λοιπόν που βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να σα παρουσιάσουμε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικέ για τη UNICEF σε όλους τους ε, τομείς μας, ε, όχι μόνο ε, για τη δουλειά μας τα παιδιά, βεβαίως ε, ασχολούμαστε με ζητήματα που αφορούν τα παιδιά και τις, τις φυσικές καταστροφές. Υιοθετήθηκαν σε υψηλό επίπεδο στην UNESCO και όλοι οι φορείς και οι οργανισμοί του ΟΗΕ συμμετείχαν ε, στην υπογραφή των κατευθυντήριων γραμμών. Ήταν μια μακρόχρονη διαδικασία που ξεκίνησε. Μας πήρε δύο χρόνια να καταλήξουμε σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, επειδή έγιναν ε, μακροσκελείς διαβουλεύσεις, βεβαίως ε, με τους εμπειρογνώμονες, αλλά και με ειδικού ε, του κλάδου. Σε 66 χώρες εργαστήκαμε και έχουμε λάβει πλήρεις ε, μελέτες από 66 χώρες. Είχαμε διαβουλεύσεις ε, σε και ελέγχου και δοκιμές στην Αιθιοπία, στο Ομαλή, Σομαλία, αναρρύθμιτες χώρες. Και θέλουμε να δούμε και να σιγουρευτούμε ότι αυτές οι κριτήρες γραμμές μπορούν να εφαρμοστούν από όλες αυτές τις χώρες αποτελεσματικά. Το κοινό στόχος μας ήταν όλες οι κοινότητες ε, και φορείς ανθρωπιστικής δράσης ε, που δραστηριοποιούνται σε τέτοιες περιοχές σύγκρουσης για να προλάβουμε και να μετριάσουμε ε, αυτά τα φαινόμενα σε όλους τους τομείς της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης δεν είναι δηλαδή μόνο για τους ειδικού του κλάδου, ε, αλλά και μη ειδικού για να καταπολεμήσουμε την ε, βία με βάση το φύλλο. Πολλά επιμέρους στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Πρέπει να οικοδομήσουμε την ε, ανθεκτικότητα με τους εθνικούς εταίρους, να στηρίξουμε τη διακυβέρνηση για να αποτρέψουμε και να καταπολεμήσουμε την βία με βάση το φύλλο. Ένα κύριο στοιχείο εδώ είναι ότι δεν προσπαθούμε μόνο να προβλέψουμε τα στοιχεία και πολύ συχνά είναι πολύ αδύναμα τα συστήματα για την παρακολούθηση και στήριξη των θυμάτων και έτσι τελικά δεν έχουμε τα στοιχεία που απαιτούνται. Υπάρχουν λοιπόν κάποια επιμέρους ε, κατακαιρματισμένα στοιχεία, αλλά δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα. Αυτό συνέβη στο Πακιστάν κατά τη διάρκεια των πλημμύρων, στο Μάλι, όπου έχουμε συγκεκριμένα φαινόμενα, όπως και στη Λιβερία. Όλα αυτά όμως είναι μη εμπεριστατωμένα. Αλλά για να αποτρέψουμε την βία με βάση το φύλλο και να βοηθήσουμε και τα θύματα, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τι έχει αλλάξει σε σχέση με άλλες κατευθυντήριες γραμμές από την Διοργανική Επιτροπή. Έχει πολύ ευρύτερο φάσμα. Ε, είχαμε ασχοληθεί μόνο με το πεδίο σύγκρουση και την αύξηση της σεξουαλικής βίας. Αυτό αποτελεί και πάλι προτεραιότητα. Όμως τώρα εξετάζουμε ευρύτερα το θέμα τη ε, βίας με βάση το φύλλο, για παράδειγμα πορνεία, ε, αναγκαστική γάμη παιδιών, εμπορία γυναικών και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα στοιχεία τα λάβουμε υπόψη σε ό,τι αφορά τη σεξιστική βία επί του περιεχομένου. Για να σας δώσω μια εικόνα του περιεχομένου των κατευθυντήριων γραμμών, εξετάζουμε τις ανάγκες διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων, διαφορετικές ε, ηλικιακές ομάδες, άτομα με αναπηρίες, ΛΟΑΔΜ, διαφορετικές αδυναμίες ή ευαισθησίες που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο της βίας Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία για την πρόληψη και αντιμετώπιση ε, της εξαιστικής βίας ό,τι αφορά την υγεία, τη διατροφή. Αναφερόμαστε σε δύο διαφορετικές κατηγορίες καταστροφών, σε αστικό και μη αστικό ε, περιβάλλον, στην Ήπεθρο δηλαδή, και όλα αυτά πώς εντάσσονται στην, στον ανθρωπιστικό κύκλο. Δηλαδή κάθε πρόταση έχει ένα συγκεκριμένο κατάλογο στοιχείων που εξετάζουμε. Για παράδειγμα, ε, πρόσφατος στο σεισμό στο Νεπάλ ή στις Φιλιππίνες, στους τυφώνες πέρυσι, είχαμε τεράστια αύξηση της εμπορίας ε, γυναικών σε τέτοιες ε, περιστάσεις φυσικών καταστροφών, αλλά και στις περιοχές συγκρούσεων, στις εμπόλεμες ζώνες δηλαδή. Όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών αρχών, λαμβάνουμε υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και παρέχεται έτσι ένα διεθνές πλαίσιο αντιμετώπισης της εξιστικής βίας. Επίσης, προσπαθούμε να υποβάλουμε case studies και να δώσουμε παραδείγματα. Πολύ σημαντικό είναι να καταφέρουμε να πείσουμε τις ε, χώρες να αναλάβουν πραγματικά και να δώσουν μεγάλη προτεραιότητα σε αυτά τα στοιχεία αυτά τα προβλήματα, τα φαινόμενα, για να αντιμετωπίσουν και να αυξήσουν την πρόληψη τέτοιων φαινομένων. Απαιτείται βεβαίως, πέραν των ειδικών και των εμπειρογνωμόνων, να υπάρχει ε, γενική κατανόηση του φαινομένου και από τους μη ειδικούς. Να υπάρχουν δηλαδή ευρείες παραπομπές ε, ε, στις καθητήρες γραμμές μας. Οι δείκτες και η παρακολούθηση, πολύ σημαντικά στοιχεία αυτά. Είδαμε λοιπόν ότι δύσκολα μπορεί κανείς ε, να δείξει τα στοιχεία σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση της στοιχής βίας ε, στον προγραμματισμό μας. Δηλαδή, να διασφαλίσουμε ότι η παρακολούθηση αυτού του ζητήματος ε, όχι απλώς συμβαίνει, αλλά και θα συνεχίσει να συμβαίνει στο μέλλον. Το πλαίσιο που προτείνουμε εξετάζει τα αποτελέσματα με βάση τις παρεμβάσεις ε, στις πληθυσμικές κατηγορίες. Βλέπουμε δηλαδή και την ε, πορεία των ε, προγραμμάτων και μπορούμε έτσι να μετρήσουμε και την πρόοδο με βάση τους στόχους μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο και θέλαμε να το επισημάνουμε και αυτό, γιατί θεωρούμε ότι αυτό θα κάνει τη διαφορά με την πάρδα του χρόνου. Τώρα, εν συντομία, να σας δώσω ένα παράδειγμα για το πώς ένας κλάδος μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη και τη μετώπιση της σεξιστικής βίας. Ο τομέας της ε, επιστημιστικής ασφάλειας πολύ συχνά συνδέεται με αυτά τα φαινόμενα. Πολύ συχνά δεν εξετάζουμε όλους τους κινδύνους σε όλους αυτούς τους κλάδους. Για παράδειγμα, η επιστηστική ανασφάλεια μπορεί να οδηγήσει σε καταναγκαστικούς ε, ή πρόωρους γάμους. Αυτό βλέπουμε τώρα στη Συρία. Ε, δίνεται προτεραιότητα στη διατροφή των αγοριών έναντι των κοριτσιών. άλλη διάσταση. Τα κορίτσια και οι γυναίκες είναι υπεύθυνε για τη διατροφή και αυτό πολύ συχνά οδηγεί σε εντάσει στην οικογένεια και υπάρχει κίνδυνος εξιστικής βία. Μετά στο Νότιο Σουδάν, για παράδειγμα, σε, μία, σε έναν από τους καταβλισμούς, τα κορίτσια φεύγουν για να μαζέψουν σιτηρά και εκεί πέρα για πέφτουν θύματα βιασμού, για παράδειγμα. Αν πρέπει να, να φύγουν μακριά από το σπίτι τους τα κορίτσια για να πάνε στο σχολείο και πάλι ε, ενδεχομένως να δεχθούν επίθεση στον δρόμο. Μετά η κατανομή του φαγητού. Πρέπει να εξετάζουμε ακριβώς πώς εφαρμόζουμε τα προγράμματά μας. Ακόμα και αν το δοχείο είναι πολύ μεγάλο, δεν μπορεί να το κουβαλήσει η γυναίκα, μπορεί να δεχθεί επίθεση. Ή αν η μάρκα φαίνεται πάνω στο δοχείο, ακόμα και αυτά τα στοιχεία. Δεν θέλω να τα αναφέρω όλα, όμως αυτά είναι κάποια παραδείγματα συστάσεων που αναφέρουμε, ούτω ώστε οι επικεφαλείς των προγραμμάτων να τα εξετάσουν αυτά τα στοιχεία για να μετριάσουν τον κίνδυνο, να αυξήσουν την επικοινωνία και αν ε, ε, αντιμετωπίσουν, εντοπίσουν μάλλον τέτοια φαινόμενα και περιστατικά να μπορέσουν να τα κοινοποιήσουν για να υπάρξει κάποιο είδους αντιμετώπιση. Τέλος, Ήδη δύο χρόνια ασχολούμαστε με αυτές τις κριτήρες γραμμές, όμως και πάλι βρισκόμαστε μόνο στην αρχή. Υπάρχει τώρα μία στρατηγική εφαρμογής και σκοπός είναι να υπάρχει κατάλληλος προγραμματισμός σε όλα τα στάδια αντιμετώπιση μιας φυσικής καταστροφής, ούτως ώστε να, να μειώνεται ο κίνδυνος, ε, να αυξάνεται η ανθεκτικότητα και να καταπολεμάται ο κίνδυνος της εξωτικής βίας. Έχουμε τρεις ε, κύριους ε, στόχους. Η συνεργασία εδώ και τώρα για να αυξήσουμε και να προβάλλουμε περισσότερο αυτή μας τη στρατηγική. Θέλουμε δηλαδή ε, κάποιους που να προβάλλουν προς τα έξω και την πολιτική μας. Ε, θέλουμε εταίρους. Δεύτερος στόχος είναι η υποστήριξη, πώς θα γίνει αυτή η εφαρμογή, πώς θα αυξήσουμε τις δυνατότητες των ανθρώπων αυτών. Τρίτος στόχος, ε, να προσελκύσουμε και χορηγούς, να συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία. προβολή αυτών των στοιχείων, ούτως ώστε να υπάρξει και συνέργεια μεταξύ ε, κυβερνήσεων και τέταρτων παρακολούθηση, εκμάθηση και αξιολόγηση, ούτως ώστε να μην μένουμε πίσω. Τελευταία διαφάνεια, αυτή τη ε, διαδικασία ε, αυτή τη στιγμή, έχουμε ξεκινήσει από τον Ιανουάριο, έχουμε και μια ομάδα εφαρμογής Συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία, συνεχίζουμε να μαθαίνουμε και ελπίζουμε να καταρτήσουμε και έναν κατάλογο παραδειγμάτων ε, που θα στελεχώσουν περαιτέρω την πρότασή μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Λιούις. Πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία σας. Και μας μεταφέρετε στην πραγματικότητα μας ενημερώνετε για τους τρόπους έμπρακτης εφαρμογής όλων αυτών των θεμάτων. Τώρα η κυρία Φλόρικα Φινκ Όιερ θα λάβει το λόγο, που είναι διευθύντρια της πολιτικής στρατηγικής και διεθνούς συνεργασίας του προγράμματος ΕΚΟ. Έχετε κι εσείς 7 λεπτά. Thank you very much. And I Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ για να υποστηρίξω με σας και με την ΤΕΒΕ τη δουλειά της UNICEF. Γιατί και εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτή την υπόθεση. Είμαστε συνεργάτες στο Είμαστε συνεργάτες στην αντιμετώπιση της σεξιστικής βίας. Υπάρχουν ε, πολλές περισσότερες συγκρούς και καταστραφές από ό,τι κατά παρελθόν και αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια, όχι όμως μόνο αυτές, αλλά και τα αγόρια έχουν να αντιμετωπίσουν ε, τη σεξιστική βία. Ακούσαμε από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής ΔΕΒΕ ότι αυξάνεται η γκάμα των βίων ε, εκδηλώσεων αλλά και έντασή τους και από ό,τι φαίνεται ε, πολλοί ασχολούνται με τον πόλεμο, με εμπόλεμες καταστάσεις, με συγκρούσεις. Ε, αλλά η βία δεν περιορίζεται μόνο στον πόλεμο και παράλληλα ε, βλέπουμε ότι και στην τρομοκρατία η σεξιστική βία χρησιμοποιείται και ως μια μορφή τρομοκρατίας και αποσταθεροποίησης. Εξάλλου, θέλω να πω ότι στηρίζουμε ανεπιφύλακτα όλη αυτή τη δουλειά, γιατί ο στόχος είναι να προκύψει μία κοινή έννοια. Ε, κοινή με την έννοια ότι θα αφορά τους δωρητές, ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γενική Διεύθυνση από την οποία προέρχομαι, αλλά και τις ε, κυβερνήσεις όλοι πρέπει, οφείλουν να εφαρμόζουν κάποιες προδιαγραφές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει σχέση με την αποτελεσματικότητα. Η Λούις ε, σας έδωσε κάποια ιδέα. Επίσης ε, αυτό που έχει σημασία είναι το πώς ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τη βία και αυτό αυτό μπορεί να γίνεται και στην ψηφιστική βοήθεια στον σχεδιασμό αυτής. Αυτό που παίζει ρόλο επίσης είναι ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρχές. Γι' αυτό εμείς ε, θέλουμε να προάγουμε ε, τις ε, κοινέ προδιαγραφές. Αυτό θα γίνει του χρόνου. Θα έχουμε μια παγκόσμια συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών και χαίρομαι πάρα πολύ που αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στις ε, μετρήσεις γιατί πιστεύω ότι ε, μόνο εάν μπορέσει κανείς ε, να κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις, μόνο και έτσι μπορεί να κάνει σωστή χρήση κονδυλίων, κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τους δωρητές αν και το βασικό θέμα θα πρέπει ε, να είναι ότι οφείλουμε να ε, δούμε λιγάκι τα οικονομικά. Έτσι λοιπόν εμείς ε, στηρίζουμε την, αυτές τις κατευθυντικές γραμμές και αυτό δεν είναι τυχαίο γιατί και από πλευρά Ηνωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς προτείνουμε μια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη της τη διάσταση του φύλου. Ε, αυτό δεν είναι απλά ως ένα έγγραφο το οποίο θα μπει στο αρχείο, αλλά ως ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θέλουμε και εμείς να ενταχθούμε και να μετρηθούμε και όπου επιτιμούμε να μετρηθούν και οι εταίροι μας. Θεωρώ ότι αυτό έχει τη σημασία του. Επίσης, θέλουμε να εξετάζεται η διάσταση του φύλου και η σεξιστική βοήθεια ε, με τρεις ε, στόχους ε, και θα ήθελα πολύ σύντομα για να γίνουν όλα αυτά πιο κατανοητά να σας αναφέρω και τρία συγκεκριμένα παραδείγματα. Αν δούμε λιγάκι στοχευμένες δράσεις, ας πάρουμε την περίπτωση του Μπαγκλαντές. Αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες, όπως η Παππούα Νέα Γουινέα, παραδείγματος χάρη. Πολλές γυναίκες ε, στο Μπαγκλαντές, το 87% των γυναικών υφίσταται οικιακή βία και όταν βγαίνουν έξω ε, αντιμετωπίζουν και πάλι βία και διάφορες ε, μορφές ε, διακριτικής μεταχείρισης, βιασμό, επιθέσεις, ε, ξαναγκασμένη εργασία, σεξουαλική εκμετάλλευση. Αυτά όλα αυξάνονται. Κατόπιν τούτου, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν στοχευμένες ενέργειες για να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αλλά και να προσφέρεται και μεγαλύτερη προστασία σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών. Μπορεί κανείς να διαφωνεί επ' αυτού, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια μορφή δράσης που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αν δούμε λιγάκι τώρα άλλες ε, βασικές δράσεις, στην Αιθιοπία παραδείγματος χάρη, ε, υπάρχει το παράδειγμα της προστασίας και, του νερού. Οποτεδήποτε προσφέρεται η υγειονομική βοήθεια, αυτό που έχει σημασία είναι να μην δημιουργείται ένα επικίνδυνο περιβάλλον ούτε για, τα γυναί για τις γυναίκες ούτε για τα αγόρια. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την κρίση στη Συρία. 18 ε, εκατομμύρια στοχευμένες δράσεις, μάλλον 18 εκατομμύρια ε, δαπανώνται για στοχευμένες ε, δράσεις ε, χρησιμοποιούνται και εκταμιεύονται από τη UNICEF και από τιμικές επιτροπές, αλλά γενικά έχουν εκταμιευτεί 33 εκατομμύρια για την αντιμετώπιση των θυμάτων της βίας, ε, της κρίσης ε, στη Συρία. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ΔΕΒΕ έχει αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα πρέπει να προσφέρεται ειδική βοήθεια στις γυναίκες και στα κορίτσια έτσι ώστε να μην εξαναγκάζονται σε ε, πολύ πρόωρους ε, γάμους που κατ' ουσίαν αυτό τι είναι, είναι ε, μία μορφή πορνείας. Επίσης, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και να στηρίξουμε περισσότερο τα προσόντα, γιατί πρέπει κανείς να διασφαλίσει Θα πω κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων ε, που βελτιώνει τις ε, δυνατότητες ε, για να μην υπάρξει εξιστική βία έναν οικιακού προσωπικού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί νομίζω ότι πρέπει στην πράξη να εφαρμόζει κανείς και αυτά τα οποία διακηρύσει. Έχουμε και κάτι το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να το συζητήσει κανείς με την πιο ευαίσθητη ομάδα που είναι οι γυναίκες και τα κορίτσια έτσι ώστε κατά την εφαρμογή όλα αυτά ε, να δοκιμάζονται αν πραγματικά βγάζουν νόημα. Κάνουμε λοιπόν τις απαραίτητες μετρήσεις. Και θα τελειώσω με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα γιατί έχουμε και συναδέλφους ε, που θα μπορούσαν και εκείνοι να μιλήσουν για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι ο συντονισμός και η συνεργασία με τους στρατιωτικούς. Ξέρετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολλές στρατιωτικές αποστολές και θέλω να σας εξηγήσω μία στο Μαλί όπου εμείς ε, πήγαμε ε, στους συναδέλφους μας και τους είπαμε θα πρέπει να διασφαλίσετε ε, στην σύλληψη της ιδέας και των ιδεών που εφαρμόζεται στην πράξη, να έχετε κατά νου και το θέμα της διάστασης του φύλου. Να υπάρχουν σχετικοί μηχανισμοί, αλλά να υπάρχει και ένας κώδικας συμπεριφοράς που οι δυνάμεις ε, στο Μαλί πρέπει να τον σέβονται. Αλλά να υπάρχει και ένας μηχανισμός λογοδοσίας. Αυτά είναι παραδείγματα ότι μπορεί κανείς να δει τα θέματα κάτω από διαφορετική γωνία. Βεβαίως όλα αυτά είναι σημαντικά ε, για μας ε, για να προσφέρουμε βοήθεια. Και μερικές φορές είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνει κανείς και επί τόπου. Αυτά είχα να πω και μπορούμε μετά αν να συζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σιέτς και Στένεκερ που εκπροσωπεί το Ταμείο για τον Πληθυσμό των Ηνωμένων Εθνών. Παρακαλώ 5 με 7 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ακούγοντας ε, τις προηγούμενες ομιλήτριες, σκεφτόμουν ότι η αναθεώρηση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, ή μάλλον γιατί οι αρχικές ήταν από το 2005. Σκεφτόμουν ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο από το 2005. Πριν από 10 χρόνια, όλος ο τομέας αυτής της εξιστικής βίας ήταν ε, μία ειδική υποκατηγορία για τους ε, εμπειρογνώμονες. Όμως δεν υπήρχε γενικό ενδιαφέρον της κοινή γνώμης για αυτό το ζήτημα. Επομένω αυτό είναι πολύ θετική εξέλιξη. Σε αυτά τα 10 χρόνια πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν αυξήσει ε, την ενασχόλησή τους με αυτό το ζήτημα και ο ΙΕ έχει ασχοληθεί πολύ συγκεκριμένα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας βεβαίως έχει υπερψηφίσει πολύ σημαντικά ψηφίσματα που προωθούν μία πιο εύρωστη ανταπόκριση στη σεξιστική βία και πολλοί νέοι πλέον επιλέγουν αυτόν τον τομέα ε, για τη σταδιοδρομία τους. Γιατί η UNFPA είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία και προτεραιότητα ε, και από μόνο του στοιχείο, αλλά και στο πλαίσιο του έργου μας ε, στην, ε, σε ό,τι αφορά την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, την ενδυνάμωση και χειρεφέτηση των γυναικών, ακόμα και τη διασφάλιση καλύτερων στοιχείων, πληθυσμιακών στοιχείων, για να έχουμε καλύτερες πολιτικές με βάση επιστημονικά στοιχεία. Έχουμε αυξήσει τις δυνατότητές μας για την ανταπόκριση της εξαιστικής βίας και σε συνεργασία ε, με την DG ECO πριν από μερικά χρόνια. Όλα τα γραφεία μας έχουν εμπειρογνώμονες για αυτό το στοιχείο και ουσιαστικά έχουμε αντίστοιχου μηχανισμούς σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε. Το 2005 με την πρώτη εφαρμογή αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών έχουν λάβει πλέον τη μορφή ενός εγχειριδίου για τους εμπειρογνώμονες, αλλά και για όλους όσοι προσπαθούσαν κάπως να παρέμβουν σε αυτόν τον κλάδο πέραν των παραδοσιακών σφαίρων, σφαίρων επιρροής. Όμως ε, μεταγενέστερες ε, αξιολογήσεις έδειξαν ότι από τις πλέον ε, στοιχειώδεις ενέργειες που είχαν προταθεί δεν εφαρμόζονται και έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος των γυναικών και των κοριτσιών δεν λάμβανε υπόψη τους ε, πολύ συγκεκριμένους κινδύνους που αντιμετωπίζουν ε, τα κορίτσια και οι γυναίκες. Πρέπει να αναφέρουμε ότι οι κατευθύνες γραμμές που έχουν τώρα ήταν αποτέλεσμα μακροσκελέστατων εργασιών δύο ετών μεταξύ UNICEF και UNFPA που ήταν επικεφαλής της διαδικασίας, αλλά και μια task force 16 οργανώσεων, οργανισμών ε, του OEA, UNHCR, UN Women, UN Food Program, αλλά και όλων των υπολείπων κύριων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Oxfam, Save the Children και πολλές άλλες. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συμμετείχαμε σε αυτό το εγχείρημα και με βάση και την ισχυρή μας παρουσία επί που θεωρούμε ότι θα πρέπει να διδραματίσουμε πολύ σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών. Τώρα, σε εθνικό επίπεδο, η στρατηγική εφαρμογή που ανέφερε συνάδελφος από την UNICEF εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους εφιστάμενους μηχανισμούς συνεργασίας και τους βασικούς παράγοντες ε, που διαμορφώνουν αυτό τον μηχανισμό σε εθνικό και διεθνέ επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί οι φορεί ε, να τεθούν επικεφαλή για τη στήριξη άλλων φορέων ε, του κλάδου για την ενσωμάτωση αυτή τη διάσταση σε κάθε τομέα πολιτική. Η εφαρμογή βεβαίω έχει τον κύριο και πρωταρχικό σκοπό τα ανθρωπιστικά προγράμματα για όλες τις επίγουσες ε, ε, περιστάσεις να σχεδιάζονται σε όλους τους κλάδους τομείς και από όλα τα διαφορετικά μέρη με έναν τρόπο τους ώστε να μειώνει τον κίνδυνο, να αυξάνει την ε, ανθεκτικότητα και να δίνει βιώσιμες λύσεις στο ζήτημα της εξιστικής βίας. Ο συνολικός στόχος των κατηδύρων γραμμών είναι να επιτύχει ευρύτατες αλλαγές, ούτως ώστε ο προγραμματισμός αυτός ε, με ευαισθησία προς την διάσταση του φύλου ε, να συνεχίζεται και να λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα προγράμματα αντιμετώπισης ανθρωπιστικών ή φυσικών καταστροφών. Όλα αυτά θα βοηθήσουν και θα βελτιώσουν σημαντικά την ασφάλεια και την ευημερία αυτών των γυναικών και κοριτσιών. Μία ενέργεια που θα μπορούσε να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ρεαλιστική μια τέτοια πρόταση, αλλά ενδεχομένω θα μπορούσε να την εξετάσει, όλοι οι εταίροι που συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόζουν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Για παράδειγμα, να ενσωματωθεί στον ε, δίκτυ, το gender marker που αναφέρθηκε προηγουμένως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Οι κατευθύντηρε γραμμές από μόνος τους δεν φτάνουν, πρέπει να εφαρμοστούν, αλλά αυτό θα ήταν ένα καλό στοιχείο. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ζεύκα Πέτκοβα, που είναι σύμβουλος στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας, ε, ειδικευμένη ε, στα θέματα ισότητας φύλων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Για πέντε λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την τις δύο επιτροπές των γυναικών και της ανάπτυξης για την οργάνωση αυτή τη ανταλλαγή απόψεων και του ευχαριστώ για τη δέσμευσή του υπέρ τη ισότητα των δύο φύλων. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση εκό, για την στενή συνεργασία που είχαμε στα θέματα προώθηση ισότητα φύλων. Αλλά να ευχαριστήσω και τη UNICEF και το UNFPA για την αργότερη προσπάθεια στην αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών. Πέντε λεπτά είναι πολύ λίγος χρόνος. Θα εστιαστώ σε θέματα σεξουαλικής σεξιστικής βίας, ε, ε, σε θέματα εμβόλεμων ζωνών και κυρίως ε, από εξωτερική άποψη, εξωτερικές πολιτικές. Καταρχήν, το 2003 είχαμε την έκκληση για ανάληψη δράση από την ΕΚΟ με πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου. Παρακολουθήσαμε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία ως σημαντική εταίρη. Και είπατε εκπρόσωπος και ειδικοί εκπρόσωποι για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής που έγινε πέρυσι στο Λονδίνο για να σταματήσει η σεξουαλική βία στις εμπόλεμες σειράξεις. Επίσης ζητήσαμε να σταματήσει η ατιμορρησία των ενόχων αυτών των εγκλημάτων. Μετά τη Σύνοδο Κορυφής του Λονδίνου, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέταξε ένα άτυπο έγγραφο, ένα οδηγό έμπρακτης δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να σταματήσει η σεξουαλική βία σε εμπόλεμες ζώνες. Πολύ περιεκτικό έγγραφο και περιλαμβάνει πολλούς τομείς. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανταπόκριση κρίση, την πρόληψη των κρίσεων και φυσικά την ανθρωπιστική βοήθεια. Ακούσαμε συγκεκριμένα παραδείγματα προηγουμένως για στρατηγική και πολιτική συνεργασία και τι κάνουμε στις αποστολές ε, ΚΕΠΑ επιτόπου. Πάντως συμφωνήσαμε και η ΕΕΔ ξεκίνησε ε, την κατάρτιση μιας μελέτης ε, με θέμα το πώς αντιμετωπίζεται η σεξιστική και σεξουαλική, σεξουαλική βία σε όλες τις αποστολές ΚΕΠΑ. Το 2015 έχουμε την επέτειο του ψηφίσματος του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, για τις γυναίκες, την ασφάλεια και την ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ανέκαθεν ε, υπέρμαχος ε, και θερμός υποστηρικτής αυτού του προγράμματος. Μάλιστα συμμετείχαμε και σε διαβουλεύσεις για την παγκόσμια μελέτη που θα γίνει φέτος για το θέμα αυτό. Και αυτή η παγκόσμια μελέτη και η παγκόσμια αναθεώρηση που θα λάβει η χώρα τον Οκτώβριο είναι σημαντικά ορόσημα για όλους μας, προκειμένου να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και να δούμε τις νέες τάσεις. Με, με τις ε, τροπολογίες στο ψήφισμα 1325 του 2013 που μιλούσε για ε, τη σεξιστική βία, είναι σημαντικό να δούμε πώς ε, λειτουργεί και το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έχουμε την περικτική και σφαιρική προσέγγιση που αναλύει την ε, εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Ένωση του ψηφίσματος 1325 και μάλιστα αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να εξυγχρονίσουμε και να επικαιροποιήσουμε τους δείκτες μας για να βελτιώσουμε την παρακολούθηση και την σωστή εφαρμογή του προγράμματος για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Γιατί πριν από 15 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, δεν είχαμε δείκτες για τη σεξιστική βία. Σήμερα έχουμε και αυτό και ο σχετικός ε, τομέας θα βελτιωθεί. Επίσης, ε, στην αναθεώρηση του Οκτωβρίου, η Ισπανία θα προεδρεύσει το Συμβούλιο Ασφαλείας και ε- η ΕΕΔ έχει στενή συνεργασία με την Ισπανία για να εφαρμοστεί αυτή η νέα σφαιρική προσέγγιση που είναι πραγματικά περιεκτική και να εμπλέκει και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο έπακρο. Ένας από τους τομείς που είναι επίση σημαντική. Καταρχήν μίλησα πριν για το ανεπίσημο αυτό έγγραφο, το non-paper, αλλά το τελευταίο μου λεπτό θα ήθελα να το αφιερώσω σε δύο έγγραφα πολιτικής ε, που εκπονούνται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και λαμβάνουν υπόψη την 20η επέτειο της πλατφόρμας του Πεκίνου ε, και την ε, δράση για την αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015. Έχουμε καταρχήν το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Εκεί η σεξουαλική βία σε εμπόλεμε ζώνε και η σεξιστική βία συμπεριλαμβάνονται, καθώς και η εφαρμογή κατευθυντηρίων γραμμών για, από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Όλα αυτά περιλαμβάνονται και επίσης ελπίζουμε το Συμβούλιο του Ιουλίου να υιοθετήσει το σχετικό σχέδιο δράση. Ένα άλλο σημαντικό έγγραφο πολιτικής που βρίσκεται υπό επεξεργασία αυτή τη στιγμή μετά τα περσινά συμπεράσματα του Συμβουλίου είναι το σχέδιο δράσης για τα φύλλα. Ε, αρχικά επικεντρωνόταν μόνο στην αναπτυξιακή μας βοήθεια. Τώρα έχουμε δέσμευση και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τη ΥΠΑ της εκπροσώπου ότι θα έχουμε ένα νέο στο στεναρό και φιλόδοξο έγγραφο που θα εξετάζει όλε τι εξωτερικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υποβάλει προτάσει για συγκεκριμένε δράσει που θα αφορούν την ανθρωπιστική ενίσχυση, αλλά θα περιλαμβάνει και συγκεκριμένου δείκτες για τη σεξουαλική βία σε εμπόλεμες ζώνες και κυρίω ε, υπό το πρίσμα της αναπτυξιακή μα ατζέντα μετά το 2015. Βάζω τελεία εδώ και περιμένω τι ερωτήσει σα. Σας ευχαριστώ. Πριν περάσουμε στη συζήτηση, και δεδομένου ότι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης ε, θα χρειαστεί να φύγει νωρίτερα από το τέλος συζήτηση, θα ήθελα να του δώσω πρώτα το λόγο ε, για να μας παρουσιάσει τα σχόλιά του μετά τις ομιλίες που ακούσαμε. Έχετε το λόγο κύριε Κούλογλου. Uh, Ευχαριστώ. Έχω ένα ερώτημα προς την κυρία Κλωρίνκα νομίζω το όνομά σας. Είπατε ότι πρέπει να συμπαριλάβουμε και τα θύματα της τρομοκρατίας. Τι εννοείται ακριβώς με αυτό. Θέλετε να απαντήσω απευθείας, ναι, αν μπορείτε. Λοιπόν, είτε πρόκειται για ένα θύμα σεξιστικής βίας, εξαιτία ενδοκογυναικής βίας, ε, εγκλήματος πολέμου, τρομοκρατίας, όπως και να έχει παραμένει ένα έγκλημα η σεξουαλική αυτή βία. Ίσως δεν ήμουν αρκετά σαφής. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στο παρελθόν επικεντρωνόμασταν ε, πάρα πολύ στην ε, σύμβαση της Γενέβης και λέγαμε ότι είναι έγκλημα πολέμου. Τώρα πλέον έχουμε νέα σενάρια που δεν εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο πια. Αν δείτε την πόκο χαράμ τον ISIS ε, και άλλες τέτοιες οργανώσεις, έχουμε αύξηση του βιασμού, της σεξιστικής βίας ως μέσο τρομοκρατίας και αποσταθεροποίησης. Γι' αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι ακόμα πιο σημαντικό πλέον, γιατί δεν λέμε μόνο ποιος ήταν ο θήτης, εξετάζουμε και το θύμα. Ε, επικεντρωνόμαστε περισσότερο στον επιζώντα δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτές τις ευάλωτε ομάδες, ανεξάρτητα από το ποιος έχει διαπράξει το έγκλημα. Όμως υφίσταται ζήτημα, πρέπει να το παραδεχθούμε. Στην περίπτωση των εκτοπιστέντων, λοιπόν, έχουμε όλα αυτά τα κορίτσια που βιάστηκαν από την Πόκο Χαράμ, επιστρέφουν στον καταβλισμό, ε, ελπίζουμε να τις έχουμε να έχουν διασωθεί. Είναι όμως μια πραγματικότητα πλέον, την οποία δεν μπορούμε ε, να αγνοήσουμε. Γι' αυτό δυστυχώς, και το τονίζω δυστυχώς, έχουν γίνει ακόμα πιο σημαντικές αυτές τις κατηγορίες γραμμές. Ο κύριος Κούλογλου, ευχαριστώ να πω δύο λόγια μόνο. Εκ μέρου της Επιτροπής Ανάπτυξης, χαιρετίζουμε τις ε, παρεμβάσεις σας σε αυτή τη συζήτηση για ένα θέμα που μας είναι ιδιαίτερα προσφυλές. Μετά το καλοκαίρι θα συζητήσουμε στο, στην Επιτροπή μας την αναθεώρηση της ε, δομής της ανθρωπιστικής βοήθειας. Εν και της Συνόδου Τη ανθρωπιστική που θα γίνει το Μάιο του 2016. Βεβαίω, και οι δικέ σα παρεμβάσεις ε, είναι ευπρόσδεκτες και στο πλαίσιο της συζήτηση που θα κάνουμε στην Επιτροπή μου. Λοιπόν, θα πρέπει να αποχωρήσω για να παρευρεθώ σε άλλη Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε. Ε, Σας ευχαριστούμε. Θα περάσουμε τώρα στη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους για να υποβάλουν ερωτήσεις. Πρώτα στην εισηγήτριά μας για το θέμα αυτό, στην κυρία Άννη Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πω ότι είναι περίεργο ότι εκείνοι οι οποίοι είναι οι πιο αδύναμοι και οι οποίοι πρέπει να προστατευτούν περισσότερο από όλου σε περίπτωση πολέμου, ε, σε περίπτωση καταστροφής, ακριβώς εκείνοι είναι αυτοί που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι. Με άλλα λόγια δηλαδή, έχουμε πλέον ένα όπλο το οποίο ε, χρησιμοποιείται σε περίπτωση καταστροφής. Πρόσφατα, ε, τώρα μόλις έγινε ο λόγος ε, για το τι ακριβώς κάνει η Μπόκο Χαράμ, πώς εκμεταλλεύεται τα κορίτσια. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε περίπτωση καταστροφής, σε συγκρουσιασικές ε, καταστάσεις, σε περίπτωση σεισμών, καταποντισμών, τα κορίτσια και οι γυναίκες εκτίθενται στη βία. Και όλα αυτά μπορεί κανείς και να τα συνδέσει και με την οικονομική κρίση στην Ευρώπη. Δηλαδή διαπιστώνουμε ότι ε, όταν υπάρχει οικονομική κρίση οι πλέον αδύναμοι εκτίθενται σε προβλήματα. Είχα αρκετά ερωτήματα να υποβάλω, τα περισσότερα όμως έχουν υποβληθεί. Ε, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το εξής, ότι η δική μας η κοινωνία, οι δικοί μας ε, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει τουλάχιστον να έχουν την απαραίτητη παιδεία. Και νομίζω ότι αυτό ελέγχθηκε από το βήμα. Το δικό μας το προσωπικό, οι άνθρωποι που τους στέλνουμε, αυτοί πρέπει να έχουν την κατάλληλη παιδεία και να γνωρίζουν πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει την ε, ε, βία, τη σεξιστική βία. Ε, τι όμως το εξής ε, ερώτημα τι είδου απαιτήσει ε, έχουμε έναντι της κυβέρνησης. Όταν δηλαδή καταβάλλονται προσπάθειες ε, για να αντιμετωπιστεί η σεξιστική βία. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, πληροφορίες που μας δώσατε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όλες αυτές. Κυρία Νόσλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μία ερώτηση πολύ συγκεκριμένα όσον αφορά τους δράστες, αλλά όσον αφορά και τα θύματα, θύτες και θύματα. Όσον αφορά τους θύτες, το ακούσαμε ότι θύτες ε, μπορεί να είναι σε μία εμπόλυμη κατάσταση, ε, οι επιτιθέμενοι, κάποιος μίλησε και για τους τρομοκράτες. Υπάρχει όμως και μία άλλη ομάδα θύτων και αυτή αν θέλετε, είναι οι άντρες ε, που ζουν σε καταβλισμούς μαζί με τις γυναίκες ε, δεν βρίσκω τα καλά λόγια να τα χρησιμοποιήσω, αλλά μπάστε να πω το εξή, ότι όταν γίνεται μια καταστροφή πάνε όλοι μέσα σε ένα καταβλισμό και βία μπορεί να ασκηθεί και μέσα στον καταβλισμό, όχι μόνο απ' έξω. Με ενδιαφέρει λοιπόν ε, να ξέρω τι γίνεται με αυτούς τους ε, θύτες και θέλω να γνωρίζω μήπως υπάρχει περίπτωση και αυτοί που προσφέρουν βοήθεια να είναι θύτες γιατί γνωρίζουμε ότι πολύ συχνά αυτοί που βοηθούν, η παιδαγωγή αν θέλετε στα σχολεία, οι εκπαιδευτές και αυτοί μπορεί να είναι θύτες. Και θα ήθελα λιγάκι να συζητήσουμε για αυτές τις ε, τρεις μορφές θητών και να κάνουμε και μία διαφοροποίηση στα θύματα. Προφανώς και υπάρχουν γυναίκες οι οποίες γίνονται θύματα ε, στις χώρες προέλευσης, της ε, πατρίδας τους. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει και πώς μετατρέπονται σε θύματα γυναίκες που μεταβαίνουν επιτόπου για να βοηθήσουν και προσφέρουν βοήθειες ε, ως ε, νοσοκόμες, ως εκπαιδευτικοί ε, και αντί παρότι αυτές θέλουν, όπως σας είπα, να βοηθήσουν, τελικά καταλήγουν να γίνονται θύματα. Έτσι, αυτή η οπτική γωνία όλων των προβλημάτων θα με ενδιαφέρε πολύ να τη συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ. Το λόγο και ο κύριος Σεμπαστιά. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ παρόμοια ερώτηση με αυτή της προλαλήσεως σας, της κυρίας Νόεχλ. Σύντομη και σαφής ερώτηση. Τι κάνουμε εμείς που έχουμε την ευθύνη για την σεξιστική βία όταν προκαλείται από τις δίθεν ανθρωπιστικές παρεμβάσεις. Ξέρουμε ότι οι στρατιώτες των Ηνωμένων Εθνών εξανάγκασαν γυναίκες σε πορνεία σε ζώνες που δραστηριοποιούνται και μερικές φορές ε, οι ίδιοι οι στρατιώτες ε, των Ηνωμένων Εθνών ε, ήταν η υπέτη για βιασμούς και άσκηση βίας. Δεν πρέπει να επικεντρωθούμε και στα θέματα διαπαιδαγώγησης των στρατιωτών. Γιατί αν δεν διορθώσουμε τα πράγματα στον οίκο μας, θα χάσουμε οποιοδήποτε οποιοδήποτε ηθικό παράστημα για να δίνουμε μαθήματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάρτ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ από την αρχή, αλλά σε συμπίπτουν οι συνεδριάσεις και είναι δύσκολο έτσι να προεβρεθούμε σε όλες. Είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό το θέμα. Κατά τύχη μάλιστα, όταν επέστρεψα στον Εμμένο Βασίλειο την περισμένη εβδομάδα, πέτυχα έναν γνωστό μου που, με τον οποίο συνεργαζόμουν στο παρελθόν, τον κύριο Σέπερντ, που ακριβώς ε, ασχολείται με αυτό το θέμα, μία γνωστή μου, συγγνώμη, ε, ασχολείται με αυτό το θέμα και προετοίμαζε λοιπόν μία κατάρτιση προετοιμασίας, ακριβώς για να μπορέσει να παρέχει φροντίδα στα θύματα επιτόπου. Και αυτό πάλι μας ε, επιστρέφει σε αυτό το ζήτημα, το πώς θα φροντίσουμε αυτούς που θα φροντίσουν μετά τα θύματα. Γιατί επιλέγουμε βέβαια τα κατάλληλα άτομα για να παράσχουν αυτή την φροντίδα και περίθαλψη, όμως και εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε αυτά τα άτομα. Ποιο συγκεκριμένα μου ανέφερε την ανησυχία της για την κατάσταση στη Συρία και ότι δεν μπορούμε να παρεύουμε καθόλου εκεί για αυτή την ε, καταστροφική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, που ούτε καν τα γνωρίζουμε απευθείας, αλλά ξέρουμε τι συμβαίνει υπογείως. Και θα Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά για πολλά χρόνια και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρές ψυχολογικές ε, συνέπειες ε, ε, των όσων συνέβησαν σε αυτές τις γυναίκες. Δύο στοιχεία ακόμα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε περιπτώσεις όπου ξέρουμε ότι κάποια πράγματα έχουν γίνει, αλλά δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει εγώ λοιπόν απέστειλα επιστολή στην ύπατη εκπρόσωπο για τους μαζικούς βιασμούς στον Ταρφούρ το περασμένο φθινόπωρο. Από όσο γνωρίζω, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι από τότε, αλλά από όσο γνωρίζω εγώ, ακόμα δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση από του επιμέρου οργανισμού. Και νομίζω ότι υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση εδώ. Όταν κάτι έχει γίνει, έχει καταγραφεί ε, και προβληθεί και από τον τύπο, αξιόπιστο τύπο και ακόμα δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση, τι συμβαίνει. Γιατί και η Σουδανή πρόσφυγα μου ζήτησε να προβάλλω αυτό το θέμα και εμεί έχουμε καθήκον να απαντήσουμε εν γέρο, ούτω ώστε οι θήτε με κάποιον τρόπο ε, να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης και εκ μέρου και των Ευρωπαίων πολιτών, ω εκπρόσωπο των Ευρωπαίων πολιτών, όταν θέτουμε ερωτήματα θα πρέπει να λαμβάνουμε και απαντήσει. Κάτι ακόμα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο κίνημα κατά της βίας εναντίον γυναικών και παιδιών, είναι η αντιμετώπιση μας σε σχέση με τα άτομα που είναι αυτόπτες μάρτυρες, αν θέλετε, αυτή, αυτής της βίας. Πολύ συχνά αυτοί οι μάρτυρες δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν θέλουν να παρέμβουν. Όμως, στον Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθούμε πραγματικά να παροτρύνουμε αυτούς τους μάρτυρες να είναι πιο ενεργοί, ε, να καταγγέλουν τέτοιου είδους περιστατικά. Αυτό συμβαίνει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα στον Τάραμ, για παράδειγμα. Εξετάζουμε αυτό το ζήτημα στη Σκωτία και θα ήθελα να δω πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα ερευνητικά προγράμματα που αφορούν πιο γενικά την βία κατά των γυναικών, πώς θα τα αξιοποιήσουμε στο δικό μας πλαίσιο. Γιατί υπάρχουν γυναίκες που παρακολουθούν και γνωρίζουν ότι άλλες γυναίκες επέφτουν θύματα βιασμού σε εμπόλεμες ζώνες. Πώς μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε και για τα σχόλια και για τις ερωτήσεις σας θα έλεγα να δώσω το λόγο στις καλεσμένες μας με αντίστροφη σειρά αυτή τη φορά και να δώσουμε ένα δίλεπτο στην καθεμία για να απαντήσει και να σχολιάσει. Πρώτα η κυρία Ζήφκα Πέτκοβα από την ΕΙΕΔ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις σας. Και εγώ να ξεκινήσω από το τέλος. Δεν ξέρω τι συμβαίνει ακριβώ με αυτή την επιστολή που αναφέρατε προ την υποτέκη αλλά θα το διερευνήσω περαιτέρω όταν επιστρέψω στην υπηρεσία μου. Θα λάβετε λοιπόν απάντηση. Για το ερώτημα του κυρίου Σεβάστια, αν όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις ε, βίας από τι δικέ μας ε, ειρηνευτικές αποστολέ, ή στρατιωτικές αποστολέ του ΟΗΕ. Αυτό είναι ένα θέμα που παρακολουθούμε εκ του συνεγγύς και στο, σε ό,τι αφορά την καταγραφή και υποβολή εκθέσεων στο 1325 ψήφισμα. Αν δείτε, υπάρχει πολύ συγκεκριμένη υποβολή εκθέσεων για το κατά πόσο και στο πλαίσιο των δικών μας αποστολών και επιχειρήσεων υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Ε, το παρακολουθούμε λοιπόν πολύ συγκεκριμένα και πολύ σοβαρά. Είπατε ποια είναι η λύση. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η κατάρτιση. Δεν μιλάμε μόνο για την κατάρτιση πριν την ανάπτυξη της επιχείρησης, αλλά και να εξηγήσουμε το φαινόμενο, τι σημαίνει, πότε συμβαίνει, πώς μπορούμε να το αποτρέψουμε. Συνεργαζόμαστε και με γυναίκες αξιωματούχους του ΟΗΕ που έχουν έρθει, αλλά και με τον ΝΑΤΟ, γιατί και εκείνοι είχαν τέτοια κρούσματα στο παρελθόν. Είναι ένας από τους τομείς που μας απασχολούν λοιπόν και έτσι το συνδέω και με άλλο ερώτημα της κυρία Χέτ για την κατάρτιση. Να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Προστασίας και Ασφάλειας και Άμυνας ε, εξετάζει πολύ συγκεκριμένα αυτές τις επιχειρήσεις και πολιτικές και στρατιωτικές. Η ευθύνη είναι το και η αρμοδιότητα είναι των κρατών μελών. Όμως, όλα και περισσότερο εξετάζουμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ε, συνοχή ε, και την ευθυγράμμιση, αν θέλετε, σε αυτή την κατάρτιση πριν την αναχώρηση, με γνώμονα τα παιδιά, τις γυναίκες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτοί είναι οι τρεις άξονες και όλα αυτά θα τα μοιραστούμε με, τα, όλα τα κρατημέλη. Έχουμε και μια σουηδική ακαδημία ε, που θα οριστικοποιήσει πολύ συγκεκριμένη κατάρτιση για τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διάσταση του φύλου. Θα μείνω εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Στένεκερ τώρα από το Ταμείο Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να απαντήσω εν συντομία στην ερώτηση του κυρίου Σεμπαστιά. Έχουμε ένα, πάντα τον κίνδυνο κάποιο μέλος του προσωπικού ή κάποιος στρατιώτης ε, ε, που ανήκει σε αποστολή διαφύλαξη της ειρήνης να είναι ο ίδιος υπέτειος αυτούργός ε, ενός τέτοιου εγκλήματος. Και είχαμε και δύστιχες καταγγελίες ε, για τη Λιβυρία και την Αϊτή από προσωπικό που συμμετείχε σε αποστολή ε, διατήρηση της ειρήνης. Οπότε συμφωνώ με την κυρία Πέτκοβα, πολύ σημαντική κατάρτιση, διαπαιδαγώγηση πριν την ανάπτυξη, αλλά και δεντολογικού κώδικες, μηχανισμοί ελέγχου, εποπτεία και φυσικά σωστή αντιμετώπιση των αυτούργων. Ευχαριστώ. Η κυρία Φλόρικα Φιν Όγερ από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Ευχαριστώ. Για το θέμα της ατιμορρησίας που επισημάνθηκε από πολλούς από ανθρωπιστική άποψη, εμείς προσπαθούμε καταρχήν να καταγγείλουμε, να ενημερώσουμε ε, βέβαια, δεν είμαστε πολιτικοί, αλλά έχουμε υποχρέωση ενημέρωσης ε, και καταγγελίας ε, και μερικές φορές υφιστάμεθα και τις συνέπειες. Και μάλιστα περιλήφθηκε πια στο πρόγραμμα των Αποστολών ΚΕΠΑ και κώδικας συμπεριφοράς, κατάρτιση, διαπαιδαγώγηση πριν την ανάπτυξη και εποπτεία, σωστός έλεγχος. Γιατί θέλουμε και σε επίπεδο πρόληψη να δράσουμε. Είναι σημαντικό αυτό για τους φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας. Τώρα, για το αν γίνεται διάκριση μεταξύ των αυτοργών και των θυμάτων. Βέβαια, εγώ σας μίλησα πολύ περιεκτικά προηγουμένως, πολύ επιγραμματικά συγγνώμη και οικογενειακή βία, αναγκαστική γάμη προς πορνεία, παρενόχληση, ε, είτε λαμβάνουν χώρα σε πόλεμο, σε πολεμική σύραξη, είτε αλλού, ε, θα πρέπει να τη χάνει μεταχείριση. Και μιλούμε για την ευπάθεια των θυμάτων. Δεν γίνεται διάκριση αν το θύμα είναι κορίτσι, αγόρι, άνδρας ή γυναίκα. Το θέμα είναι, υπάρχει κίνδυνος για μεγαλύτερη έκθεση σε βία υπάρχει ενισχυμένος κίνδυνος και αν ναι, πώς θα προσπαθήσουμε να μετριάσουμε αυτή την τροτότητα των θυμάτων. Δεν κάνουμε λοιπόν διάκριση ούτε μεταξύ αυτούργων, ούτε μεταξύ θυμάτων. Έχουμε μερικές φορές στοχευμένες δράσεις, οι γενικές δράσεις, αλλά ακόμη και οι γενικές δράσεις ε, ελέγχονται με μηχανισμούς συμμόρφωσης και με δείκτες και εξετάζουμε τις ιδιαιτερότητες ε, ιδιαίτερα όταν υπάρχει υψηλός ή ενισχυμένος βαθμός έκθεσης και αύξηση της τροτότητας, ευπάθειας. Τώρα, διάλογος με την ΤΠΚΟ, με επικεφαλή στην ΕΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί συμμετέχουμε στο διάλογο αυτό και προσωπικά ήμουν παρούσα πολλές φορές και φυσικά υψώνουμε και τη φωνή μας, ανοχή μηδέν, αλλά το θέμα είναι να μην μείνουμε στα λόγια, να περάσουμε στα έργα και φυσικά να δούμε και τόπου πώς ε, ε, λειτουργεί το σύστημα, πώς εφαρμόζεται και να ενημερώνουμε. Φυσικά ε, ο κόσμος έχει γίνει επικίνδυνο μέρος για όλους και για το προσωπικό ανθρωπιστικής βοήθειας. Και το θέμα της πρόσβασης, το θέμα της προστασίας, του σεβασμού του ρόλου των, του προσωπικού ανθρωπιστικής βοήθειας. Η προσέγγιση δυστυχώς ε, δεν είναι σωστή. Δεν υπάρχει ο ούτε από πλευράς κυβερνήσεων, ούτε από ένοπλες δυνάμεις. Και η παροχή ανθρωπιστική βοήθειας γίνεται όλο και πιο δύσκολη και χαίρομαι που το επισημάνατε, γιατί θα πρέπει και εμείς ε, να βρούμε άλλους μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και φυσικά οι εταίροι μας θα πρέπει να εξετάσουν και αυτό το θέμα. Γιατί εμείς είμαστε δωρητές αλλά και είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε βοήθεια, αλλά πολλές φορές η πρόσβασή μας είναι δύσκολη. Πάντως με, μέσω των εταίρων μας υπάρχει πρόσβαση στη Συρία. Εκεί οι εταίροι μας με κίνδυνο τη ζωή τους πραγματικά παρέχουν αξιέπαινες και αξιοθαύμαστες υπηρεσίες και το κάνουν καθημερινά. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τέλος η κυρία Γκουίν Λιούις από τη uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να αναφερθώ σε αυτά που έχουν ήδη λεχθεί και να υπογραμμίσω το γεγονός ότι σε κάθε σύγκρουση έχουμε και διαφορετικές, διάφορες μορφές ε, επιζώντων αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι ότι ε, πρέπει να αποφύγουμε εκ των προτέρων της ε, κατηγοριοποίησης, να δούμε το πώς μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Θέλω επίσης ε, να αναφέρω και το πλαίσιο που έχουμε, δηλαδή είναι η προστασία από την σεξουαλική εκμετάλλευση και τις καταχρήσεις. Υπάρχουν οι διεθνείς ΙΜΚΟ και ο στόχος είναι να προσφέρουμε ε, στους ε, εργαζόμενους ε, που είναι αντικείμενο σε την προστασία. Αυτό βεβαίως έχει και σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές για τους ΛΟΑΔ αλλά ο κύριος Σίνκ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής, θέλω να σας πω ότι είναι μια πολύ ενεργός ομάδα κατά την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών. Ε, στόχος είναι, όπως σας είπα, να μπορούμε να διασφαλίσουμε όλες αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές οπουδήποτε ενεργοποιούμεθα. Βεβαίως ε, και όλοι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι ανεξάρτητα με το που εργάζεται κανείς, σε ποιο τομέα, τι είδους ευθύνη φέρει ε, ο καθένας ε, για να μπορεί να διασφαλίσει ότι υπάρχει ένα δίκαιο σύστημα για όσους επιζούν. Όλοι μας έχουμε ένα ρόλο να διαδραματίσουμε. Νομίζω ότι υπάρχει η σωστή φιλοσοφία ως προς το τι προσπαθούμε να προάγουμε και στη Συρία σας είπα είμαστε παρόντος, η UNICEF, ο ειδικό Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών εκεί έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια πρόκληση και νομίζω ότι εφαρμόζουμε ε, πολύ σημαντικά προγράμματα, πραγματικά προσπαθούμε να προάγουμε την ε, προστασία και να έχουμε πρόσβαση να πλησιάσουμε τα πιο ε, ευαίσθητα και τροτά θύματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τους προσκεκλημένους μας. Είναι μια συζήτηση που θα τη συνεχίσουμε και στην Επιτροπή των Γυναικών. Κάποια συμπεράσματα που θα μπορούσαμε να αντιλήσουμε είναι καταρχήν η σημασία ε, εφαρμογής, ε, συντονισμού, αξιολόγησης ε, και εποπτείας αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, καταμέτρησης αυτών των, της εφαρμογής αυτών των κατευθυντήριων γραμμών και καταπολέμηση όχι μόνο της σεξουαλικής βίας αλλά και της εξιστικής βίας σε όλες τους τις εκφάνσεις. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παράγοντες επιδείνωσης του κινδύνου και να λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές πτυχές της πραγματικότητας ε, σε κάθε τομέα. Επίσης, στη στρατηγική αυτή είναι σημαντικό να αναμίξουμε, να εμπλέξουμε τις γυναίκες και τις ε, ομάδες ιδιαίτερου κινδύνου. Πολύ χρήσιμη κατά τη γνώμη μου η συζήτηση. Όπως σας είπα δεν θα μείνει εδώ, θα συνεχιστεί στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για την συμβολή σας. aliás. Muito eh, Περνάμε τώρα στο σημείο 8 της σημερινής διάταξης. Συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2016 και εντολή για τον τριμερή διάλογο. Η Επιτροπή μας αποφάσισε να συντάξει γνωμοδότηση επί της έκθεσης της Επιτροπής Προϋπολογισμών με θέμα την εντολή για τον τριμερή διάλογο για τον προϋπολογισμό του 2016. Η συγγήτρια της γνωμοδότησης, η συντάκτρια μάλλον της γνωμοδότησης, είναι η κυρία Ματέρα από το ΕΛΚ. Τη γνωμοδότηση της ήδη τη συζητήσαμε στη συνεδρίαση της 7ης Μαΐου και είχαμε προθεσμία μέχρι τις 18 Μαΐου ε, για την κατάθεση των τροπολογιών. Κατατέθηκαν συνολικά 11 τροπολογίες στη γνωμοδότηση. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι θα συζητήσουμε αυτές τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για τη γνωμοδότηση Ματέρα και θα ψηφίσουμε επί της γνωμοδοτήσεως αύριο το πρωί. Κυρία Ματέρα που αλλά την αντικαθιστά η κυρία Πετήρ που θα μας παρουσιάσει τη θέση της συντάκτηρας της γνωμοδότησης. Παρακαλώ, κυρία Πετήρ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Ματέρα που δυστυχώς κολλείεται για λόγους υγείας να έρθει στη συνεδρίαση. Το όνομά της είναι αναπόσπαστα δεμένο με την γνωμοδότηση αυτή. Μόνο 11 τροπολογίες, όπως είπατε, κατατέθηκαν στην γνωμοδότηση της κυρίας Ματέρα. Και έχοντας υπόψη ότι το έγγραφο της Επιτροπής με τις προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνει ε, ισορροπημένα στοιχεία σε ό,τι αφορά την ισότητα των δύο φύλων, Γι' αυτό η κυρία Ματέρα εξέφρασε την δυσαρέσκειά της και κάλεσε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν για να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική στρατηγική που στο μέλλον και στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς θα λάβει υπόψη και την ισότητα των φύλων. Επίσης η κυρία Ματέρα επισημαίνει ότι και προσωπικά ίδια αλλά και η ομάδα του ΕΛΚΑ θέλει να αυξηθούν στον προϋπολογισμό ημνίες θεμάτων γυναικών και ισότητας των δύο φύλων. Και γι' αυτό η κυρία Ματέρα συμφωνεί σχεδόν με όλες τις τροπολογίες που κατέθηκαν από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Από την άλλη πλευρά, η συγγήτρια είναι κατά τις τροπολογίες της κυρίας Μπιόρκ, τις τροπολογίες Περθών 10, Βέβαια, εκτιμά την ε, συνεισφορά της κυρίας Μπιόρκ και της ομάδας Γκουε, αλλά θεωρεί ότι η τροπολογία 10 είναι υπερβολικά τραβηγμένη και ακατάλληλη για τη γραμματότηση. Μάλιστα, στην τροπολογία αυτή καλούνται τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, τις στρατιωτικές δαπάνες. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καν προπολογισμό για στρατιωτικέ δαπάνε. Οπότε είναι τελείω ανεδαφική η σχετική τροπολογία. Είναι εκτό θέματο. Η κυρία Μπιόρκ ζητά μείωση των στρατιωτικών δαπανών και ανακατεύθυνση των δαπανών αυτών σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Το θέμα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, η ε, ιδιαίτερη τροπολογία αυτή είναι δεν γίνεται δεκτή. Είμαστε κατά στο ΕΛΚ, αλλά επαναλαμβάνω, είναι και αναδαφική τροπολογία επειδή δεν υπάρχει καν στρατιωτικό προπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν στρατιωτικέ δαπάνε. Πάντω η κυρία Ματέρα είναι κατά τη τροπολογία 10, ζητά να την καταψηφίσετε. Κατά του λοιπού είναι υπέρ των υπόλοιπων τροπολογιών και σα καλεί να υπερψηφίσετε τη γνωμοδότηση αύριο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο κύριε Ρέντκε από τους Πράσινους. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ αντικαθιστώ την Μόνικα Βάνων, ε, τη συνάδελφό μου, που ε, δεν μπορούσε να έρθει, αλλά ε, θέλω να πω μερικά πράγματα και θέλω να σας πω ότι θέλω να ευχαριστώ και εγώ και εκ μέρους του αδέλφου μου την εισηγήτρια για τη γνωμοδότησή της. Αποτελεί μια πολύ καλή βάση για περαιτέρω συζητήσεις και υπάρχουν κάποια σημεία που η κυρία Βάνα θέλει να συζητήσει, να τονίσει στη συζήτηση. Ε, αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη βία κατά των γυναικών. Αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα. Εμείς ως πράσινοι ε, προφανώς υποστηρίζουμε ότι η βία κατά των γυναικών πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα. Ε, επίσης, αυτό που θέλω να αναφερθεί είναι η οικονομική κατάσταση των γυναικών. Παραδείγματος χάρη, ε, το ότι υπάρχει διαφορά στις αποδοχές και αυτό πρέπει να το λάβει κανείς υπόψη του και από δημοσιονομική σκοπιά. Άρα δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημασία της βίας ε, κατά των γυναικών, αλλά υπάρχει και το οικονομικό θέμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Κατόπιν, έχει συντάξει την τροπολογία υπαριθμών 2, όπου θέλει να ενισχύσει το ρόλο του δημόσιου τομέα για τις ε, γυναίκες. Ε, πολλές γυναίκες εργάζονται στο δημόσιο τομέα, από την άλλη όμως ε, και οι παροχές του δημοσιοτομέα είναι πολύ σημαντικές για τις ε, γυναίκες. Ε, επίσης να πούμε ότι αυτό δεν καθίσταται πλέον απόλυτα σαφές, άρα δηλαδή θα ήθελε να υπάρχουν και τα δύο αυτά στοιχεία στον δημόσιο τομέα και να συμπεριληφθούν στη γνωμοδότηση. Σε γενικές γραμμές πρέπει να σας πω, είμαστε ευχαριστημένοι με αυτή τη γνωμοδότηση και αν αυτό ε, γίνει αποδεκτό, νομίζω ότι η σκιώδη εισηγήτρια από τη δική μας ομάδα θα χαρεί ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Από τους σοσιαλιστές ε, και δημοκράτες ε, δίνω το λόγο στη σκιώδη εισηγήτρια την κυρία Μπόρζαν. Χωρίς μικρόφωνο κυρία Μπόρζαν. Θεωρώ ότι η χειραφέτηση των γυναικών ε, δεν μπορεί να λάβει χώρα χωρίς την οικονομική τους ε, χειραφέτηση. Και φυσικά η ενίσχυση των κοινωνικών δικτύων για να γίνει δυνατός ο συνδυασμός προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Ε. Και είναι σημαντικός αυτός ο στόχος. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτε είναι υπέρ τη πλειοψηφίας των τροπολογιών και θα θέλαμε να, να ευχαριστήσουμε τη συντάκτηρα της γνωμοδότησης. Ευτυχώς αποσιάζει, αλλά θα σας το μεταφέρετε. Είχαμε θαυμάσια συνεργασία και να ευχαριστήσω ιδιαίτερως και τη γραμματεία. Θεωρώ ότι θα καταφέρουμε με τη συμφωνία μας να ενισχύσουμε την ε, τυχή αυτή των γυναικών και τη συμπερίληψή τους ε, και τη θεματισότητα των φίλων στον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Eh, Σας ευχαριστώ. Εγώ θα μιλήσω εκ μέρους ομάδας μου, μια και απουσιάζει και ο δισηγητριά μας. Θα ήθελα να πω ότι είναι προφανές πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δική της στρατιωτική δύναμη, δεν έχει δικό της στρατό αλλά έχει πολλές δαπάνες για το συντονισμό των στρατιωτικών δυνάμεων, ιδιαίτερα σε εξωτερικές της παρεμβάσεις. Οπότε είναι αλήθεια ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός, μια και χρηματοδοτεί την ΕΙΕΔ, έμεσα χρηματοδοτεί και στρατιωτικά θέματα. Και το είδαμε και προηγουμένως. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να εστιαστούμε και να αφιερώσουμε περισσότερα κονδύλια στο θέμα της ισότητας των φύλων, περικόπτοντας δαπάνες που γίνονται αλλού. Και γι' αυτό σας καλώ να υπερψηφίσετε την σχετική τροπολογία, την υπαριθμό 10 της ΓΚΟΕ. Δεν ζήτησε άλλος κανείς το λόγο. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Πετήρ αν επιθυμεί να δευτερολογήσει. Όχι. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση και περνάμε στο σημείο 10 της της διάταξης που έχει θέμα το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020. Πρόκειται για γνωμοδότηση που θα υποβληθεί στην έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής ΕΜΚΟ, της Επιτροπής Απασχόλησης. Έχουμε δει το σχέδιο γνωμοδότησης ε, της συντάκτριας ε, της κυρίας Μπίλιανα Μπόρζαν από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και σήμερα θα έχουμε την πρώτη συζήτηση επί του σχεδίου γνωμοδότησης. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην εισηγητριά μας, τη συντάκτρια της γνωμοδότησης μάλλον, στην κυρία Μπίλιανα Μπόρζαν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε το θέμα αυτό σήμερα, γιατί κατά τη γνώμη μου πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την αγορά εργασίας. Εγώ από την επαγγελματική μου εμπειρία ε, ως γιατρός ε, σε θέματα εργασίας. Ε, ξέρω πως ε, η εργασία υπό δυσμενείς συνθήκες επηρεάζει την σωματική αλλά και την ψυχική υγεία. Και οι συνθήκες εργασίας μερικές φορές επηρεάζουν την ίδια τη φυσιογνωμία των γυναικών και έχουν σχέση και με τις υποχρεώσει που έχουν οι γυναίκες και στο σπίτι, γιατί το ωράριο εργασία των γυναικών δεν σταματάει ε, στην εργασία τους, στην απασχόλησή του, στο χώρο απασχόλησης, αλλά συνεχίζεται στο σπίτι με άλλη μορφή. Γι' αυτό λοιπόν ε, ε, εκφράζω τη θλίψη μου για την ανάκληση της οδηγίας για, τις, για άδεια μετρότητα και επίση ε, το θέμα τη έκθεση σε επικίνδυνε ε, τοξικέ ουσίε. Ακόμη δεν έχει αναφέρει ε, δεσμευτικά όρια έκθεση για τον για μεγαλύτερο αριθμό τοξικών ουσιών. Επίση, μιλούμε για την αύξηση του αριθμού των μειοσκελετικών παθήσεων μεταξύ των γυναικών που απορρέουν από τι συνθήκε εργασία. Δυστυχώ, επειδή έχουμε περιορισμό στην έκταση τη γνωμοδότησης, δεν μπόρεσα να περιλαβώ όλα τα στοιχεία που θα ήθελα να συντάξω, αλλά θα υποβάλω και εγώ τροπολογίες και σας καλώ να κάνετε και εσείς το ίδιο για να διαβρύνουμε τη γνωμοδότηση. Επίσης, ε, θα ήθελα να ασχοληθώ με τις γυναίκες που εργάζονται στον ιδιωτικό χώρο των ε, πελατών, αλλά και στις μετανάστριες. Επίσης, να επιστήσω την προσοχή στο θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης και του στρες που υφίστανται εξαιτία των βραχυπρόθεσμων συμβάσεων εργασία ή της ε, χαμηλής, χαμηλότερης ομοιβής σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους. Επίσης θα πρέπει να προβλέψουμε και για τις γυναίκες κατάλληλη ιατρική ε, περίθαλψη και περίθαλψη υγείας. Θα πρέπει να περιλάβουμε τη διάσταση του φύλου στα θέματα αξιολόγηση του κινδύνου. Ε, θέλουμε ίση μεταχείριση σε θέματα αυτά, στην πρόσβαση στην υγεία. Και επίσης ε, ε φαίνεται φαίνονται διαφορές και από τις διαφορές στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ ανδρών και γυναικών και μεταξύ κρατών μελών. Είναι εντυπωσιακέ αυτές οι διαφορές μεταξύ των χωρών μελών εξαιτίας της άνης πρόσβασης που, υπάρχουν, που υπάρχει στην υγεία. Αυτά και παρακαλώ να συνεισφέρετε με τις τροπολογίες σας για να βελτιώσουμε τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία εισηγήτρια. Δεν ζήτησε κανείς το λόγο. Εγώ σκιώδη εισηγήτρια της GUNGL. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για την γνωμοδότησή σας. Γενικώ συμφωνώ με όλες τις ιδέες της γνωμοδότησής σας. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε στην γνωμοδότηση. Είναι προφανές όμως ότι εξαιτία ε, του περιορισμού της ε, έκτασης ε, δεν μπορέσετε να εμβαθύνετε στα επιμέρους θέματα. Χάρη στις όμως θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στην γνωμοδότηση και να την εμπλουτίσουμε. Ένα από τα θέματα που μας ανησυχούν ιδιαίτερα είναι η αύξηση του, των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στο χώρο εργασίας η αύξηση των ψυχικών ασθενειών στον εργασιακό χώρο, που πλήττουν περισσότερο τις γυναίκες. Ε, επίσης, η ανεργία πλήττει τις γυναίκες με αποτέλεσμα να ε, αποδυναμώνει την ψυχική τους υγεία. Γιατί αυξάνονται οι πιέσεις, οι ψυχολογικές, αυξάνονται οι πιέσεις από τους εργοδότες, αυξάνεται η ένταση εργασίας σε περίπτωση που εργάζονται και ακριβώς επειδή υπάρχει μεγάλη ενέργεια και είναι δύσκολο να βρει μια γυναίκα θέση απασχόληση, υφίσταται πολύ ε, μεγαλύτερες πιέσεις και περισσότερο άγχος. Και ακριβώς επειδή είναι δύσκολο να βρουν θέση, οι γυναίκες υποβάλλονται σε συνθήκες και ανέχονται συνθήκες που προηγουμένως ήταν ε, ανεπίτρεπτες και απαράδεκτες. Και τα προβλήματα της ψυχικής υγείας ε, αυξάνονται εντυπωσιακά ενώ δεν υπάρχουν προληπτικές, ε, πολιτικές ούτε πρόληψης ούτε θεραπείας δυστυχώς για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ψυχικά προβλήματα. Καλό θα ήταν λοιπόν ε, να ληφθούν υπόψη αυτά τα προβλήματα και να αναπτυχθούν μέθοδοι για την καταπολέμησή τους και σχετικές πολιτικές και να υποβληθούν συγκεκριμένα μέτρα. Ένα άλλο θέμα αφορά τη ρύθμιση του ωραρίου εργασίας, του χρόνου εργασίας. Πολύ σημαντικό ζήτημα. Επίσης να αντισταθούμε στην απόπειρα απορρίθμισης του ωραρίου εργασίας. Γιατί η μεγάλη αντασεργασία έχει συνέπειες στην υγεία. Το αναφέρει και η συγγήτρια αυτό. Επίσης, εκεί που μιλάτε ε, για την ανταλλαγή των μέτρων των πρακτικών και την ε, κατάρτιση των επιθεωρητών εργασία. σίγουρα η κατάρτιση και η διαπαιδαγώγηση είναι πολύ σημαντικά θέματα, ιδιαίτερα για την ισότητα των δύο φύλων. Και φυσικά υπάρχουν εκπρόσωποι για την ασφάλεια και επιθεωρητές, αλλά δυστυχώς όλο και λιγότεροι. Και μπορεί στη θεωρία να υπάρχουν αυτές οι δομές, αλλά στην πράξη αυτοί οι ίδιοι επιθεωρητές προβαίνουν σε απολύσεις. Οπότε τέτοιου είδου ε, δομές καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιούνται εις βάρος των εργαζομένων ή να μην αποδυναμώνονται. Θα πρέπει να ενισχυθούν. Για όλα αυτά τα θέματα θα καταθέσουμε τροπολογίες, ευελπιστώντας ότι θα συμβάλλουμε στην έκθεση, στην διαμόρφωση της γνωμοδότησης μάλλον. Η κυρία Μούντι. Yes, just... Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα ήθελα να στηρίξω όχι μόνο την κρατική εκπροσώπηση, αλλά και την συνδικαλιστική παρέμβαση και τον ρόλο των, ε, των σωματείων σε ό,τι αφορά την ε, ασφάλεια. Και στηρίζω και τις ε, προτάσεις αυτές, ιδίως σε δύο τομείς. Πρώτον, η εργασία με βάρδιες και πιο συγκεκριμένα νυχτερινή βάρδια και οι προεκτάσεις ό,τι αφορά την υγεία των γυναικών και την ασφάλειά τους και μετά η αύξηση της απόστασης γιατί οι γυναίκες εργάζονται σε όλα και μεγαλύτερη ηλικία εξαιτία της έλλειψη ε, δυνατοτήτων συνταξιοδότηση. και αναγκάζονται να δουλεύουν για πολύ περισσότερο από αυτό που θεωρείται μια συνήθι ε, ηλικία συνταξιοδότηση. Όμως ε, είναι εξαιρετική αυτή η πρωτοβουλία και εμείς θα στηρίξουμε, εγώ δηλαδή, θα στηρίξω όσο μπορώ περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ. Ήθελα απλώς να πω ότι η κυρία Μπόρζαν έθεσε τον δάκτυλο επί των τύπων των ήλων. Αναγνώρισε τα πιο σημαντικά προβλήματα και ε, την ευχαριστώ γι' αυτό. Θα υποβάλω τροπολογίες για την οδηγία για το ωράριο εργασίας. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι μιλούμε για γυναίκες που στον τομέα των υπηρεσιών μπορεί να δουλεύουν ε, επί τρεις συναπτές εβδομάδες, δεν έχουν καθόλου χρόνο ανάπαυσης, ούτε Σαββατοκύριακο ελεύθερο και υποαμείβονται και όλα και οι περισσότερες ξεκινούν ε, από τα 16-18 να εργάζονται. Οπότε τα φτάνουν στην όριμη ηλικία. Έχουν ήδη υπονομεύσει τόσο πολύ την σωματική και ψυχική τους υγεία που είναι πραγματικά θλιβερό. Αυτό το πρόβλημα θα το επισημάνω σε τροπολογίες που θα υποβάλω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο λόγος και πάλι στην εισηγήτριά μας, στη συντάκτρια της γραμματότησης, αν θέλει να σχολιάσει τις παρατηρήσεις που άκουσα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συναδέλφους που υπέβαλαν προτάσεις. Συμφωνώ μαζί τους και σίγουρα η γνωμοδότησή μου δίνει απλώς το σκελετό θα το γεμίσουμε με τις τροπολογίες και τις προτάσεις σας. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε και ελπίζω ότι και άλλοι συνάδελφοι που σήμερα απουσιάζουν θα καταθέσουν τροπολογίες και θα εμπλουτίσουν την γνωμοδότηση. Εγώ πιστεύω ότι με τη συνεργασία θα καταλήξουμε σε πολύ θετική γνωμοδότηση που θα βοηθήσει και τους συναδέλφους ε, ε, της ε, Επιτροπής Απασχόλησης. 22 Ιουνίου να σας υπενθυμίσω ότι λύγει η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ε, η Γραμματεία με πληροφορεί ότι η η, κατάθ... η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών λήγει στις 22 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Διεκπαιρεώσαμε τη σημερινή ημερήσια διάταξη. Αύριο η συνεδρίαση ε, θα ξεκινήσει στις 10. Στις 9 θα συνεδριάσουν οι συντονιστές, 9 με 10. Αυτά για σήμερα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Χαίρετε.